Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίασή μας με την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Βλέπετε ότι θα συνεδριάσουμε μόνο το πρωί. Δεν έχουμε προγραμματίσει συνεδρίαση το απόγευμα ούτε αύριο, διότι Μεταξύ άλλων, είναι περίπλοκη η διαδικασία για τη συζήτηση για τη ΜΥΦΙΤ και το ΜΥΦΙΡ. Η διαδικασία για τη συζήτηση αυτή είναι περίπλοκη και γι' αυτό τα αφαιράσαμε ως σημεία από την ημερήσια διάταξη. Την εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ. Να σας κάνω μια ανακοίνωση. Ένας τριμερόγης διάλογος έλαβε χώρα στις 29 Φεβρουαρίου ο πρώτος και ο δεύτερος χθες για το IORP. Portfolio Transfer, Depository, Αποθετήριο Τίτλων, ε, βασικά θέματα, περιβαλλοντικά ε, κίνδυνοι για την περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβέρνηση, αξιολόγηση αντικτύπου, δεν έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για αυτή την πλειάδα θεμάτων, ωστόσο έγινε αρκετά καλή πρόοδος και μπορεί να υπάρξει συμβαστική λύση κυρίως για το αποθετήριο. Και στις 13 Απριλίου θα είναι η επόμενη συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Πάμε στο σημείο 3. Ε, εικονικά νομίσματα. Δίνω το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε τη μεγάλη χαρά να εργαστούμε πάνω σε μια νέα τεχνολογία. Την τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από το bitcoin. Πάρα πολλές είναι οι κινητομίες, η τεχνολογία κινείται ταχύτατα, είναι συναρπαστικές οι εξελίξεις και θέλω να ξεκινήσω όχι διότι έχουν τελειώσει οι διαβουλεύσεις μας για το θέμα αυτό, αλλά γιατί θεωρώ ότι οι περασμένες εβδομάδες ήταν εξαιρετικά επικοδομητικές, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι ενεπλάκησαν σε αυτές τις συζητήσεις και αυτό ισχύει και για τους συναδέλφους. Στρέφομαι προς αυτούς, διότι ασχολήθηκαν με την υπόθεση, διάβασαν το φάκελο, οι αλλαγές που κόμισαν είναι πολύ χρήσιμες κατά τη γνώμη μου και Μπορέσαμε να καλέσουμε πάρα πολλούς εμπειρογνώμονες στις ακροάσεις και εδώ ε, στη συνεδριά της Επιτροπής και να διαβουλευτούμε με αυτούς με τηλεδιάσκεψη επίσης. Και όλες αυτές οι παρουσίες, όλοι αυτοί οι ομιλήτες συνεισέφεραν τα μάλα, μάθαμε πολλά ε, και χάρη στην εξαιρετική δουλειά της αγραμματείας βεβαίως. Τα βασικά που θέλω να τονίσω είναι τα εξής. Πρώτον, δεν είναι μόνο κάτι με το οποίο ασχολούνται ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, αλλά και οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται ιδιαίτερως για το δυναμικό, της δυνατότητας αυτές της, αυτής της τεχνολογίας. Ε, πάνω από ένα δις ευρώ έχουν επενδυθεί σε αυτό το τομέα σήμερα. Ξεκίνησαν πάρα πολλές επενδύσεις σε σχέση με το ε, bitcoin καταρχάς και Σιγά σιγά έχουμε φτάσει στον τομέα της εκαθάρισης, του διακανονισμού ε, και της ε, αλυσίδα των μπλοκ σε αυτή την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, Distributed Ledger Technology. Δεν θέλουμε να παρακολούθησουμε αυτές τις καινοτομίες γιατί είναι πολλά υποσχόμενες. Έχουμε πάρα πολλά να κερδίσουμε σε επίπεδο παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας και περισσότερα από αυτού θα πω αργότερα. Όμως, συνάμα, πάρα πολύ είναι οι ενδυνάμοι κίνδυνοι που ε, δημιουργούνται, κυρίως εάν αρχίσει ξαφνικά να χρησιμοποιείται εξαιρετικά ευρέως η τεχνολογία αυτή. Επομένως, πώς θα είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε γρήγορα εάν δημιουργηθεί συστημικός κίνδυνος σε ένα επαρκές μέγεθος και σε ικανό μέγεθος να αποτελέσει πραγματικά κίνδυνο δηλαδή. Και γι' αυτό προτείνω να έχουμε μια task Force που με την εμπειρογνωμοσύνη της θα προτείνει γρήγορες αλλαγές στην νομοθεσία και θα συμβουλεύσει τα κράτη-μέλη πώς να αντιμετωπίσουν καλύτερα ε, τις προκλήσεις που ενδεχομένως προκύψουν με την ευρεία και διαδεδομένη χρήση τέτοιων τεχνολογιών στο μέλλον. Επίσης, Υπάρχει και το θέμα του ανταγωνισμού και της βιομηχανικής πολιτικής και θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στην εξέταση του θέματος. Δεν ξέρουμε πόσο ευρέως διαδεδομένη θα είναι η χρήση αυτής της τεχνολογίας σε 10 χρόνια από τώρα. Όμως, εάν πρόκειται να χρησιμοποιείται ευρέως η τεχνολογία σε 10 χρόνια από τώρα, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο θα έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να βεβαιωθούμε ότι χρησιμοποιείται δίκαια, ότι τα κυρίαρχα συστήματα ε, δεν θα είναι ιδιοκτησιακά, δεν θα μπορούν να κλείνουν τον ανταγωνισμό και να τον αποκλείουν και γι' αυτό θέλουμε ανοιχτή πρόσβαση, ψηφιακό πορτοφόλι, αλλά ενδεχομένως παρεφερείς ρυθμίσεις να είναι απαραίτητες. Προς το παρόν όμως δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις ακριβείς τεχνολογικές εξελίξεις. Η έκθεση αναφέρεται σε δύο ε, ζητήματα. Καταρχάς τα εικονικά νομίσματα αυτά κάθε αυτά. Και εκεί ε, τι λέμε. Τα εικονικά νομίσματα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά να χαμηλώσουν τα κόστη συναλλαγών, κυρίως τις διασυνοριακές συναλλαγές, που σήμερα παραμένουν αρκετά ακριβές, οφείλει να ομολογήσει κανείς. Και ε, έχει γίνει τεράστια έρευνα σε όλο αυτό το τομέα των ενταλμάτων. Οι εργαζόμενοι που στέλνουν χρήματα στις πατρίδες τους σε μικρές δόσεις σε άλλες χώρες, στις αναπτυσσόμενες χώρες και λοιπές, όπου ε, δεν έχουν όλοι τραπεζικό λογαριασμό, αυτό ε, είναι αρκετά ακριβό. Επομένως, ο συνδυασμός της με την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και αλυσίδας των μπλοκ έχει το δυναμικό πραγματικά τη δυνατότητα να χαμηλώσει, να μειώσει το, κόστο της, το κόστος της συναλλαγής. Και έτσι το κόστος πληρωμής και εξυπηρέτησης, αν θέλετε, θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό στην Ευρώπη. Όχι λόγω νέων κανονισμών, αλλά λόγω και χάρη στη νέα τεχνολογία. Και αυτά, όλα αυτά μπορούν να ενισχυθούν και ε, ε, αφορούν δραστηριότητες που καλύπτονται από την οδηγία για το ενίο σύστημα πληρωμών και το ενίο χώρο πληρωμών. Στις μικροπληρωμές, πολύ μικρές πληρωμές, ενδεχομένως είναι ενδιαφέρον να χρησιμοποιηθεί και αυτή η τεχνολογία μεταξύ άλλων, η οποία σταδιακά ε, μπορεί να αντικαταστήσει την πληρωμή για πολλές υπηρεσίες δεδομένων εταιρείε μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δικά μας προσωπικά δεδομένα, να φυλάξουν την ιδιωτική μας ζωή πολύ καλύτερα από τη στιγμή που θα έχουν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία. Βέβαια, κάθε τεχνολογία συνοδεύεται από κινδύνους. Μπορεί να υπάρξει ξέπλυμα χρήματος, φόρο διαφυγή, και σύμφωνα με πρόσφατες ευρωπαϊκές εκθέσεις μπορεί να ε, ε, υπάρξει χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Παρόλο που δεν υπάρχει κανένα στοιχείο μέχρι σήμερα ε, που υποδεικνύει του λόγου του αληθές. Το bitcoin είναι αρκετά προειδοποιητικό εδώ, γιατί αρχικά είχε θεσμοθετηθεί και δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να λειτουργεί με τον αυτόματο πιλότο. Όταν όμως προέκυψαν τεχνολογικά προβλήματα, δεν υπήρχε διαχειριστική δομή που θα έκανε τακτική ενημέρωση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για το bitcoin. Τέτοιου είδου ζητήματα λοιπόν διδασκόμαστε ότι μπορεί να προκύψουν. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα προστασίας του καταναλωτή από τη στιγμή που προκύπτουν και αναδύονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα και το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο ο κάθε ένας θα τηρήσει τις υποσχέσεις του. Και υπάρχει και το τεράστιο ζήτημα της μεταβλητότητας ε, του bitcoin και αυτό εγείρει ζητήματα προστασίας του καταναλωτή. Μακροπρόθεσμα όμως, ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι Υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού ε, σε τομείς πέραν των πληρωμών. Ο πιο, η πιο συναρπαστική χρήση είναι αυτή που μας ε, επισήμανε ένας εμπειρογνώμονος από το MIT σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ηλεκτρονικά εισιτήρια. Εάν σήμερα δηλαδή κανείς πουλά ηλεκτρονικά εισιτήρια για μια αθλητική διοργάνωση μπορεί να προσπαθήσει να τα πουλήσει πέντε φορές στην ίδια θέση, το ίδιο εισιτήριο και τελικά πέντε άνθρωποι να εμφανιστούν στο γήπεδο για την ίδια θέση, για το ίδιο εισιτήριο. Με αυτή την τεχνολογία όμως του κατανεμμένου καθολικού ενδεχομένως αυτό αποφεύγεται. Το ίδιο ισχύει και με την μουσική, η οποία ε, πωλείται ψηφιακά μέσω του διαδικτύου. Επομένως υπάρχουν πολλές και διαφορετικές χρήσεις που είναι εφικτές και δυνατές με αυτή τη τεχνολογία. Η πιο συναρπαστική όμως και αυτή που μας αφορά κυρίως είναι ε, η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού έτσι όπως χρησιμοποιείται στον τομέα των πληρωμών και κυρίως ε, στη δραστηριότητα της εκαθάρισης και του διακανονισμού μπορούμε να έχουμε δημόσια λυσίδα των μπλοκ όπου δεν χρειάζεται ξεχωριστή αρχή ρυθμιστική αλλά έχουμε και ιδιωτική αλυσίδα των μπλοκ η οποία μπορεί να κάνει συναλλαγές, υπολογισμούς και ε, συνάμα να παρέχει αρκετή επαρκή ικανοποιητική ασφάλεια. Θεωρώ ότι θα έχουμε ευρεία χρήση της τεχνολογίας αυτής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Βλέπω ότι δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα. Πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξουμε τις υποδομές για να είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε τάχιστα εάν χρειαστεί να νομοθετήσουμε και να ρυθμίσουμε γρήγορα να παρεύουμε και να είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Κύριο για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. ζητώ συγγνώμη είμαι μια ατελής, ένα ατελές υποκατάστατο του κύριου Ματουσέλου που δεν μπορεί να είναι εδώ να διαβάσω αυτά που σας γράφει πρώτον να καλωσορίσω την σημαντική αυτή έκθεση πρόκειται για ένα νέο φαινόμενο που εξελίσσεται ταχύτατα και η προσπάθεια του Κοινοβουλίου να καταλάβει το φαινόμενο αυτό και να προσπαθήσει επίσης να το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα της εξέλιξης των εικονικών νομισμάτων είναι ευπρόσδεκτο ε, βήμα. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Γιάκο Βάιτσικερ για, τις, ε, για την παρουσίασή του και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία μαζί του. Έχουν οργανωθεί από ό,τι ξέρω αρκετέ ε, συναντήσεις οδών εισηγητών που καλύπτουν πολλά σημαντικά θέματα. Στην αρχική φάση των συζητήσεων θα ήθελα να θέσω κάποια λίγα σημεία. Ένα. Ορισμοί. Για το τμήμα της ενίσχυσης της ρύθμισης για την εξασφάλιση της εκαιρότητας στο σημείο 10 το κείμενο αναφέρει ότι η βασική νομοθετησή θα εφαρμόζεται βάσει των δραστηριοτήτων που διεξάγονται. Το άλλο θέμα είναι ότι ο ορισμός στο σημείο α της έκθεσης, μάλλον το σημείο α της έκθεσης αφορά τους Θέλω να ξέρω από πού προκύπτει ο ορισμός. Πού τον βρίσκουμε. Σημείο 12 της έκθεσης. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προβληματική, διότι ο εισηγητής σαν συνιστά αναθεώρηση της νομοθεσίας της Ένωσης για τις πληρωμές. Πριν ζητήσουμε νέα νομοθετική ρύθμιση, θα ήταν σημαντικό να δούμε τι εφαρμόζεται τώρα και πώς. Να τσεκάρουμε δηλαδή κατά πόσο η υφιστάμενη νομοθεσία καλύπτει τις ανάγκες. Για ποιο λόγο θα λειτουργήσει αυτή η task force, η οριζόντια ομάδα, ομάδα Το σημείο 14. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Το σημαντικό είναι εδώ να υπογραμμιστεί η ανάγκη για μια μελέτη αντικτύπου δεδομένης και της σημασία ε, να έχουμε better regulation, ένα θέμα του Επίτροπου Τίμερμανς. Αυτές είναι οι πρώτες αντιδράσεις στην πρώτη ανάγνωση της έκθεσης στην ε, Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ. Ο κ. Φόξ για τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Φων που ανέλαβε την θέση του εισηγητή. Είναι ισορροπημένη έκθεση, αντιμετωπίζει τα βασικά θέματα των εικονικών νομισμάτων και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις νέχνες τεχνολογίες και την χρήση του. Συμφωνώ ότι με το εικονικό νόμισμα περιορίζονται οι μη θελμένες, το μη κόστη μεταβιβάσεων και βελτιώνεται η οικονομική ανάπτυξη. Συμφωνώ επίση μαζί του ότι πρέπει να ξέρουμε τον περιορισμένη, την περιορισμένη ικανότητα που έχουν οι ρυθμιστικέ αρχέ για να αντιμετωπίσουν και να προλαμβάνουν την εξέλιξη τη τεχνολογία. Μπορεί να είναι πλεονέκτημα το εικονικό νόμισμα αν δεν χρησιμοποιείται από εγκληματίες και τρομοκράτες. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι χρειαζόμαστε μια προσέγγιση νομοθετική που θα είναι αναλογική. Δεν θέλουμε αυτή την καινοτομία να την εξαντλήσουμε στην νομοθετική αντιμετώπιση ή να την ε, υπονομοθετήσουμε οδηγώντας τη στην εγκληματικότητα εικονικά νομίσματα βρίσκονται ακόμα σε νηπιακό στάδιο. Δεν θα ήθελα να επεκταθεί η νομοθεσία κατά τη, του ξεπλήματος ε, χρήματος της Ένωσης. Δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση στη φάση αυτή. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τη χρήση των εικονικών νομισμάτων πριν ε, επιδιώξουμε περαιτέρω νομοθετική αντιμετώπιση. Επίσης, δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η φυστάνομη νομοθεσία για τις πληρωμές, γιατί δεν καλύπτουν τους ορισμούς τα εικονικά νομίσματα ούτε πιστεύω ότι πρέπει να επεκτείνουμε το, τις διατάξεις της οδηγίας ε, πληρωμής υπηρεσιών στα εικονικά νομίσματα. Πιστεύω ότι έκανε κάνουν έκτημα να είναι θετικά για τους καταναλωτές και θα έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί να μην θέλουμε να νομοθετούμε επί παντός επιστητού με την πρώτη ευκαιρία. Θα παρότρινα τον εισηγητή να το κάνει να κάνει το ίδιο. Ευχαριστώ. For Κύριος Γέτζεκ για την Άλντε. Well, world... Πρόεδρε. Δύσκολος ο κόσμος των εικονικών νομισμάτων. Οι νομοθέτες έχουν την επιλογή να προτείνουν είτε ακραία μέτρα για τον έλεγχο των εικονικών νομισμάτων, είτε να μην κάνουν τίποτα και να αφήσουν τα εικονικά νομίσματα και τις ε, συνδεδεμένες με αυτά τεχνολογίες να εξελιχθούν. Η προσέγγιση πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση. Είδαμε αυτή την εβδομάδα ότι η Ρωσία εισάγει νομοθεσία που καθιστά εγκλήματα την, ε, τις συναλλαγές με bitcoin. Οι χώρες της Ένωσης ακολούθησαν διαφορετικές ε, προσεγγίσεις. Άλλες ε, εφαρμόζουν στα bitcoin ε, διατάξεις που αφορούν το ξέπλυμα χρήματος ή τη νομοθεσία για, για τις πληρωμές. Άλλοι θεωρούν ότι δεν είναι νόμισμα. Αυτό που προκύπτει από την έκθεση είναι ότι υπάρχει και δυνατότητες και κίνδυνοι που συνδέονται με την ανάπτυξή τους αυτή. Αυτό είναι θέμα που η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι ευρωπαίοι νομοθέτες θα έπρεπε να παρακολουθούν προσεκτικά. Η διασυνοριακή φύση των ε, συναλλαγών με bitcoin για παράδειγμα σημαίνει ότι μια ενοποιημένη προσέγγιση ανά την Ένωση είναι επιθυμητή. Ωστόσο, έχω την άποψη ότι κάθε νομοθετική ρύθμιση πρέπει να προτείνεται με πλήρη επίγνωση των συνεπειών της. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους, όχι όμως να ε, καταστήλουμε την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό καλωσορίζω την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριλάβει τα εικονικά νομίσματα στην νομοθεσία του ξεπλήματος ε, για χρημάτων. Η ψευδόνιμη ονομασία εικονικό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εγκληματίες για χρηματοδότηση. Δεν έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν κάτι τέτοιο προς το παρόν, παραμένει ωστόσο το ενδεχόμενο. Καταρχήν καλωσορίζω την ιδέα μιας task force για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των τεχνολογιών αυτών. Θα εξετάσουμε ποιος, ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση της task force για να εξασφαλίσουμε ότι η Ένωση θα βοηθήσει και δεν θα περιορίσει την ανάπτυξη των εφαρμογών με τρόπο που θα μεγιστοποιήσει τα πλονεκτήματα της χρήσης τους. Επίσης η Task Force θα έπρεπε να έχει υπόψη του και διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία του καταναλωτή και την προστασία δεδομένων. Κλείνω. Η έκθεση είναι στέρη βάση για να προχωρήσουμε και προσβλέπω σε περαιτέρω συζητήσεις για την, ε, μετά την υποβολή των τροπολογιών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. E, Ο Μιγγέλ Βιέγκας για την, ε, για την e. Καλημέρα. Το φαινόμενο είναι καινούριο σύνθετο, αβέβαιο. Ακούσαμε πολλά για το θέμα. Μιλούμε για κάτι που οικονομικά δεν έχει σημασία. Αν δείτε τα στοιχεία που υπάρχουν, βλέπουμε για ένα μικρό, πολύ μικρό ποσοστό εμπορίου. που υπάρχει και μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα που προκύπτουν από την προσφορά του χρήματος, τον σύνθετο χαρακτήρα αυτών των νομισμάτων και στο μέτρο που εξελίσσονται τα σύνθετα αυτά χαρακτηριστικά υπάρχουν διαδικασίες που επιτρέπουν την παρακολούθηση αυτών των νομισματικών των εικονικών νομισμάτων. Βέβαια υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με την νομιμοποίηση αυτών των ε, νομισμάτων γιατί μπορεί να υποκρύπτουν ε, εγκληματικές δραστηριότητες. Κατόπιν έχω πολλές επιφυλάξεις για, ως προς την δυνατότητα των νομισμάτων αυτών να παίξουν ένα, το βασικό νομισματικό ρόλο. Μονάδα αξίας και ανταλλαγής. Η πρόσβαση είναι δύσκολη, η περίοδος ε, επιβεβαίωσης του νομίσματος είναι εμπόδιο, δηλαδή ε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γενικευθεί. Άλλωστε μιλάμε για μικροπληρωμές. Επίσης, ε, το νόμισμα αυτό είναι εξαιρετικά ευμετάβλητο. Είδατε πώς συσχετίζεται το bitcoin και τα άλλα νομίσματα. Δεν έχει κανένα, καμία σχέση. Όταν λοιπόν Λοιπόν, μιλούμε για ένα bitcoin ως μέτρο αξίας. Καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε μακράν του να πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία αυτού του φαινομένου, την νομοθέτηση αυτού του φαινομένου, είναι προφανές ότι το σύνθετο, τα σύνθετα χαρακτηριστικά του δημιουργούν προβλήματα. Ένα από τα μεγάλα πλονεκτήματα του, των εικονικών νομισμάτων είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να περάσεις από έναν τρίτο. Ε, τράπεζα, κράτος, ε, εγγυητή, στον οποίο, τον οποίο εμπιστεύεται ο πολίτης. Χρειάζεται λοιπόν νομοθεσία, χρειάζεται προστασία του καταναλωτή, ωστόσο η προσπάθεια αυτή μπορεί να οδηγήσει σε λάθος δρόμο. Να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε κάποια δικαιώματα που δεν θα τηρούν, που δεν θα πληρούν τις εγγύσει που ανέφερα. Τούτου λεχθέντος φορολογικά και σε θέματα παράνομων δράσεων είναι προφανές ότι όσο μεγαλώνει, όσο εξελίσσεται και αν αναδεικνύεται το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες που εκφράστηκαν εδώ. Παρακολουθούμε λοιπόν τη θεματική με πολύ ενδιαφέρον και όπως κάναμε μέχρι τώρα θα συμβάλλουμε για να έχουμε ένα κείμενο που θα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Greens, Scott Thank you, Chair. Για τους πράσινους τώρα, Πολύ μου άρεσε η συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες που οργάνωσε ο εισηγητής και μάθαμε πολλά πράγματα για την αλυσίδα των μπλοκ και με... μου θύμισε τα χρόνια τα φοιτητικά. Μας αρέσει επίσης η ξεκάθαρο, ξεκάθαρος τρόπος με τον οποίο εξηγεί τα πράγματα στην εκθεσή του εισηγητής και βέβαια το ενδεχόμενο υπάρξουν και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Πάντω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει περισσότερε κατευθύνσει ό,τι αφορά τι προτεραιότητε να μην περιοριστούμε σε μια απλή περιγραφή του δυναμικού που υπάρχει στη τεχνολογία αυτή, διότι εν τέλει εκπροσωπούμε του πολίτε τη Ευρώπη και νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να δώσουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την νομοθετική δραστηριότητα που επιθυμούμε να δούμε. Για την ίδια την τεχνολογία τώρα, μας αρέσει το δυναμικό που έχει να προωθήσει την ε, συμπερίληψη όλων των ανθρώπων. Και εδώ παίζει ένα ρόλο και το λεγόμενο ηλεκτρονικό πορτοφόλι που έχει ε, σημασία γιατί πολλοί βρίσκονται μακριά από τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες. Μας ενδιαφέρει επίσης η διάκριση που κάνει ανάμεσα στη ιδιωτική σφαίρα και ανωνυμία. Είναι ενδιαφέρουσε οι ιδέες του εισηγητού για την χρήση της τεχνολογίας DLT και ιδίως για τις ε, επαφές που έχουν οι ε, πολίτες με διάφορες υπηρεσίες. Πάντως, επειδή πιστεύουμε ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας ήδη είναι υπερβολικά μεγάλος ό,τι αφορά τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι διευκολύνσεις στο κόστος των διαμέσων που θεωρούμε τους άλλους το κόστος είναι πολύ χαμηλό. Με την ευκαιρία αυτή θα συμφωνήσω με τον Ashley Fox, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, Συμφωνούμε όμως ότι η ρύθμιση δεν θα πρέπει να ε, φρενάρει την καινοτομία. Και η τεχνολογία αυτή που αναπτύσσεται μπορεί τελικά να υποφελήσει για το κοινό. Επίσης, όπως είπα και πριν, οι πράσινοι ενδιαφέρονται να διατηρηθούν τοπικά νομίσματα, τα οποία μπορούν να είναι και εικονικά, αλλά θα είναι σε περιορισμένη χρήση και για, για ορισμένα είδη συναλλαγών. Και δεν θέλουμε βέβαια οποιαδήποτε νομοθεσία να αναστείλει την πρόοδο αυτών. Αναμένουμε λοιπόν τις περαιτέρω συζητήσεις και ευχαριστούμε και πάλι τον εισηγητή για την ενδιαφέρουσα συνεργασία. Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα Κάπελ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για την πραγματικά επαγγελματική δουλειά που έχει κάνει και τις πολλές ε, συναντήσεις με εμπειρογνώμονες που οργάνωσε. Οι συνομιλίες ήταν πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και μάθαμε ε, πολλά πράγματα και ήταν μια καλή εισαγωγή στην τεχνολογία αυτή. Υπάρχουν παραπάνω από 600 ε, προγράμματα εικονικών νομισμάτων. Το bitcoin είναι το μεγαλύτερο, ε, το μερίδιο της αγοράς του είναι της τάξης του 90% και για μια συνολική αξία περίπου 5 δις ευρώ. Αυτά τα δείχνει καθαρά η έκθεση, καθώς επίσης και την τεχνολογία DLT, που είναι σημαντική όχι μόνο για τα εικονικά νομίσματα, αλλά και για πολλά άλλα. Έχουμε ήδη και μιλήσει για τον ε, τομέα FinTech. Το ίδιο για διακανονισμό και ε, συμψηφισμό και διάφορα τέτοια. Είναι επίσης πολύ σημαντικά ε, τα σχετικά για την ταυτοποίηση, ταυτότητας και περιουσιακών στοιχείων κλπ. Και η ΕΣΜΑ έχει κάνει ανάλυση τέλη Ιανουαρίου φέτος για την χρήση της DLT του κατανεμένου καθολικού, δηλαδή υπάρχουν ήδη φαντ τα οποία ασχολούνται με εικονικά νομίσματα, δύο από αυτά στην Ευρώπη. Υπάρχουν μορφές εμπορίου που ασχολούνται με αυτές και ε, το DLT, αυτή η τεχνολογία DLT θα αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Κυρίως ε, για την αγορά ε, χρεογράφων. Αξιογράφων δηλαδή θα αλλάξουν πολλά πράγματα λόγω ή χάρη στην χρήση της ε, τεχνολογίας DLT. Έρχομαι στο δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να θέσω υπόψη του εισηγητή, δηλαδή τις δυνατότητες που ανοίγει η τεχνολογία των, οικονομικών, των εικονικών νομισμάτων. Υποστηρίζω αυτά που ανοιγει η τεχνολογια των των εικονικων νομισματων υποστηριζω αυτα που λεει για την βελτίωση της ευημερίας πολλών, ότι θα μειωθεί το κόστος των ε, συναλλαγών και μέχρι μάλιστα 7% σε διαμεθοριακές συναλλαγές. Και μάλιστα ίσως το όφελο αυτό να ανέλθει μέχρι τα 20 δισεκατομμύρια πανευρωπαϊκά τον χρόνο. Πέρα από αυτό, η τεχνολογία για την ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων ε, συναλλαγών έχουν ένα τεράστιο δυναμικό, όπως είπα, στον συμψηφισμό και στους διακανονισμούς. Βέβαια υπάρχουν και μειονεκτήματα όπως λέχθηκε και ε, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η χρηματοδότηση τρομοκρατίας, δυνατότητα δηλαδή ανώνυμων μεταφορών χρηματικών ποσών και έλλειψη ενός αξιόπιστου νομικού πλαίσιου. Κάτι που μου λείπει από την έκθεση είναι ο κίνδυνος αυτού του κυβερνοεγκλήματος που βλέπουμε να αυξάνεται διαρκώς διότι όσο πιο ψηφιακές είναι οι συναλλαγές, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος του κοινωνεγκλήματος που το κόστος του εκτιμάται ήδη στα 400 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τώρα, smart ή better regulation. Λέει σωστά ο νομοθέτης ότι και οι ρυθμιστές αγγίζουν τα όρια τους πλέον, διότι η τεχνολογία κάνει άλματα προς τα εμπρός και δεν υπάρχουν πολλοί που να τα γνωρίζουν και ούτε τα δεδομένα είναι επαρκή που διαθέτουν οι ρυθμιστές. Γι' αυτό πιστεύω δεν θα πρέπει να κάνουμε νέες ρυθμίσεις όσο δεν γνωρίζουμε προς τα που κινείται η τεχνολογία. Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν στη βάση μόνο της τεχνολογίας. Επίσης, η δημιουργία μιας οριζόντιας task force στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βρίσκει επιφυλακτική θα ήθελα η task force αυτή να ιδρυθεί από την ίδια την αγορά. Εγώ βλέπω και πανεπιστήμια και επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τις τεχνολογικές εξέλιξεις και ασχολούνται πολύ με αυτές, αυτές να φτιάξουν μια task force. Θα καταθέσω δε τροπολογίες σχετικά. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για το τμήμα τώρα αυτό που το λέμε Catch the Eye, Νίνα Γκίλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ με τη σειρά μου τον εισηγητή για την έκθεση. Πολλοί συνάδελφοι τόνισαν την ανάγκη να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην νομοθετική ρύθμιση και στην ε, αποφυγή ε, τροχοπέδηση στην καινοτομία. Ε, το λέει αυτό ο εισηγητής. Λέει λοιπόν ότι η νομοθετική ρυθμίση θα πρέπει να είναι αναλογική και να μην αναχαιτήσει την ε, καινοτομία. Το σημαντικό είναι ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι αλλάζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Αν δούμε τα 12 δισεκατομμύρια που δημιούργησαν σε επενδύσεις με στα πλαίσια του Fintech και αν δούμε πώς το Apple Pay αλλάζει την προστασία του συστήματος νομίζω ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η νομοθετική ρύθμιση πρώτον δεν πρέπει να αναχαιτήσει την καινοτομία ούτε θέλουμε να την κάνουμε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό η ιδέα αυτή δημιουργία της ειδική ομάδα Task Force με εμπειρογνώμονε να προωθηθεί γρήγορα, διότι βλέπουμε τόση πολλή καινοτομία τα τελευταία 7 χρόνια και οι αλλαγέ στον χώρο αυτό είναι τόσο δραματικέ που νομίζω ότι πρέπει ε, να επιμείνουμε ώστε αυτή η ομάδα να ιδρυθεί ταχύτατα. Ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας λάβει τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Δεν έχει σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπερνομοθετήσει γύρω από τα εικονικά νομίσματα. Μας ενδιαφέρουν ωστόσο οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την ανωνυμία. Έχουμε και το σχέδιο δράσεως για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ανακοινώθηκε στις αρχές του χρόνου. Θα προτείνουμε λοιπόν συγκεκριμένες τροπολογίες για την οδηγία, για την ε, ε, αποτροπή του πλησίματος βρώμικου χρήματος και θα ζητήσουμε να φτιαχτούν πλατφόρμες ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων στην οδηγία. και θα υπάρχουν και αυτοί οι wallet providers, αυτοί οι πάροχοι δηλαδή ε, του πορτοφολίου, του ηλεκτρονικού πορτοφολίου που θα είναι κάτι σαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έχει εκδώσει ήδη εκδώσει προειδοποίηση ε, για τους κινδύνους της επένδυσης σε εικονικά νομίσματα λόγω της μεγάλης αστάθειάς τους και επιθυμώ επίσης να υπενθυμίσω ότι το bitcoin που είναι το βασικό εικονικό νόμισμα είναι σχετικά μικρή αγορά σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές σε bitcoins. Χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω, είναι στο επίπεδο καρτών ε, δώρου. Ε, ωστόσο είναι χρηματική αγορά. Για την ώρα λοιπόν δεν έχουμε σκοπό να νομοθετήσουμε, να προτείνουμε δηλαδή νομοθεσία, παρά μόνο για πολύ συγκεκριμένες πτυχές. Τώρα για την τεχνολογία DLT, δηλαδή του κατανεμμένου καθολικού, που είναι σχετικά νέα και είναι αυτή που αποτελεί τη βάση για τα εικονικά νομίσματα. Η DLT προέκυψε τον τελευταίο χρόνο. Άρχισαν οι ερευνές για να δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί ως εργαλείο για υποδομές πληρωμών. Αρχίζουν να γίνονται οι εφαρμογές αυτές. Κάνουμε και κάποιες έρευνες για την εφαρμογή της στον κόσμο των securities. Έχουν αρχίσει, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αρχίσει να ερευνά. Η πρόσκλησή σας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ιδρύσει μια ε, ειδική ομάδα, μια task force, μπορεί να λάβει συγκεκριμένη μορφή η Γενική Διεύθυνση Φυσπα και Connect συζητούν για την ίδρυση Task Force για την ψηφιακή καινοτομία. Αυτά θα τα περιλάβουμε σε πράσινη βίβλο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και, τις, ε, και την καινοτομία στις σχετικές υπηρεσίες. Η DLT λοιπόν θα αποτελέσει θέμα το οποίο αξίζει τη συγκεκριμένη προσοχή της Task Force η οποία θα ιδρυθεί σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ο εισηγητή κ. Φων Βάιτσέκερ. Έδειξε νομίζω η σημερινή συζήτηση ότι θα χρειαστεί να συνεχίσουμε η ομάδα των συναδέλφων να συζητούμε το θέμα αυτό ήταν σε συζήτηση αναμένω με ενδιαφέρον τις τροπολογίες και διακατέχομαι από κάποια αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε χρήσιμους συμβασμούς. Δύο ουσιώδη σχόλια τώρα για τις ερωτήσεις του Ντάριους Ροζάτη. Ο ορισμός προέρχεται από ε, έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν προσπαθούμε να κρύψουμε τίποτα, ούτε προσπαθούμε να προσετεριστούμε ή να ε, ε, παρουσιάσουμε σαν δικό μας τον ορισμό. Τώρα για το πού μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία αυτή, για την DLT δηλαδή, αναφέρομαι στην έκθεση της ΕΣΜΑ, που τονίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στους τομείς της ε, διατήρησης περιουσιακών στοιχείων, ε, ε, συμψηφισμού, διακανονισμών και ούτε καθεξής. Ολοκληρώνοντας, επιθυμώ να επανέλθω σε αυτή την προσπάθεια ακροβασίας σχετικά με το τι θα πρέπει να νομοθετηθεί σε ό,τι αφορά ευκαιρίες και κινδύνους. Πιο ενδιαφέρον μου φαίνεται είναι, και το τόνισαν και άλλοι συνάδελφοι, το ερώτημα πότε να προβούμε στην νομοθετική ρύθμιση. Το θέμα εδώ, και γι' αυτό στο σχέδιό μου κάνω την πρόταση να ιδρυθεί αυτή η task force, θεωρώ ότι όσο περισσότερα γνωρίζουμε ως κοινοβούλιο, ως ρυθμιστές για τα θέματα αυτά, όσο περισσότερο είμαστε σε επαφή, τόσο περισσότερο μπορούμε να περιμένουμε δεν θέλω δηλαδή να φτιάξω ένα γραφείο κρατικών τέρας, διότι σίγουρα ορισμένοι ανησυχούν για ενδεχόμενη τέτοια πρόπτικη. Η ιδέα είναι να επενδύσουμε στις ικανότητές μας, στην δυνατότητά μας μάλλον, να μπορέσουμε να αναμείνουμε λίγο περισσότερο με τη ρύθμιση, κάτι το οποίο μπορεί να αποφέρει και κάποια πλεονεκτήματα. Εάν περιμένουμε λίγο περισσότερο δηλαδή, μπορούμε να ρυθμίσουμε το θέμα καλύτερα. χωρίς να είμαστε αφελείς ωστόσο. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, τι τρέχει, τι εξελίσσεται. Αυτή είναι η ιδέα στην βάση της προτάσεως για την Task Force. Δεν έχω καμία διάθεση να ξοδέψω χρήματα των φορολογουμένων. Θα δαπανίσουμε κάποια χρήματα για να αποκτήσουμε κάτι και αυτό θα είναι η ικανότητα να γνωρίζουμε καλύτερα πότε είναι ο έκθετος χρόνος για να προβούμε στην νομοθετική ρύθμιση. Αυτό ήθελα να ε, τονίσω ως επιχείρημα. Και αναμένω βεβαίως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προτάσεις τροπολογιών σας. Ευχαριστώ πολύ. Καταληκτική προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 22 Μαρτίου το μεσημέρι, 19 Απριλίου εξέταση τροπολογιών, 25-26 Απριλίου ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια στις 2 Μαΐου. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο σημείο Τέσσερα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα. Μία από τις δύο νομοθετικές προτάσεις της δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Ιανουαρίου. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε ατυχές το γεγονός ότι το Συμβούλιο ήδη έχει φτάσει σε πολιτική συμφωνία πριν την ψήφιση της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως αυτό δεν αλλάζει το χρονοδιάγραμμα, διότι σε κάθε περίπτωση η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη. Επομένως θεωρούμε ότι υπήρξε μία περιφρόνηση του ρόλου του Κοινοβουλίου και κάτι τέτοιο δεν χρειαζόταν, πόσο μάλλον ε, που ε, θεσμικά είναι καταχυρωμένος ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Τούτων λεχθέντων δίνω το λόγο στον κύριο Ροτζάτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, η οδηγία που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η οδηγία που τροποποιεί την οδηγία 16 του 2011 για τη διοικητική συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών των κρατών μελών και αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής που συνέταξε και προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του τρέχοντος έτους. Και καλώς σημειώνεται κύριε Πρόεδρε ότι είναι πολύ ατυχές το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει ήδη υιοθετήσει πολιτική απόφαση για το ζήτημα αυτό, χωρίς να δώσει την ευκαιρία στο Κοινοβούλιο να εκφέρει την άποψή του. Αυτή η οδηγία αποφασίστηκε με τη διαδικασία της απόφασης το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχει ρόλο συμβουλευτικό. Ωστόσο, η σωστή διαδικασία θα ήταν το Συμβούλιο να περιμένει το Κοινοβούλιο να εκφέρει την άποψή του. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω στείλει επιστολή αναφερόμενος στο ζήτημα αυτό στον κύριο Ντάισελμπλουμ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Eurogroup. Και αυτή τη στιγμή έχει και την Προεδρία του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά εκφράζοντας ε, τη βαθιά μου ανησυχία για την απόφαση αυτή. Επί της ουσίας τώρα. Στόχος της οδηγίας είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών και να αυξηθεί, να ενισχυθεί η διαφάνεια σε φορολογικά θέματα μέσω της άμεσης εφαρμογής των συστάσεων του ΟΣΑ στην έκθεση ΠΕΠΣ. Είναι ένα έγγραφο αυτό, τη σύνταξη του οποίου είχαν ζητήσει οι G20 και στην 13η δράση η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μία σειρά προτύπων, στάνταρ δηλαδή, για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών. Με στόχο τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής για τις επιχειρήσεις που αποσκοπούν να ε, ε, έχουν το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς να αποφύγουν τελικά να πληρώσουν φόρους, tax planning και tax avoidance. Οι φορολογικές αρχές χρειάζονται συνολικά και περιεκτικά στοιχεία για τα οικονομικά αποτελέσματα των πολυεθνικών ομίλων και χωρίς πρόσβαση σε τέτοιου είδους στοιχεία και τέτοιου είδους πληροφορίες είναι δύσκολο να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, aggressive tax planning. Και γι' αυτό απαιτείται οι εταιρείες να υποβάλουν ετησίως τέτοιου είδους στοιχεία, να ε, υποβάλουν στις φορολογικές αρχές κάθε, χώρες, ε, κάθε χώρα στις οποίες δραστηριοποιούνται στοιχεία για διάφορες οικονομικές μεταβλητές. Έσοδα π.χ., ε, κέρδος επί των πωλήσεων προφόρων, φόρος εισοδήματος καταβληθής και ο οφειλόμενος, δηλωθέν κεφάλαιο, ε, παρακρατούμενα έσοδα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, μη διανεμηθέντα ε, κέρδη, κέρδη προφόρων και ούτω καθεξής. Και επομένως αυτομάτως και υποχρεωτικώς ανταλλάσσονται τα στοιχεία αυτά μεταξύ φορολογικών αρχών δηλαδή τα κράτη-μέλη οφείλουν να υποβάλουν τα στοιχεία σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο φορμάτ, με μια συγκεκριμένη ε, μορφή να έχουν, να έχει υποβιώλη αυτών των στοιχείων. Αυτή η υποχρέωση όμως όλο αυτό το πράγμα περιορίζεται στις εταιρείε των οποίων ο κύκλος εργασιών ξεπερνά τα 750 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Φαίνεται ψηλό αυτό το νούμερο, φαίνεται πολύ ψηλό αυτό το κατόφλι, ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το κατόφλι αυτό καλύπτεται το 90% όλων των διασυνοριακών ροών μεταξύ πολυεθνικών εταιριών και ομίλων. Επομένως καλύπτεται πραγματικά η μερίδα του λέοντος των ενδυνάμει βλαβερών, επιβλαβών αν θέλετε, φορολογικών πρακτικών από πλευράς μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η οδηγία βεβαιώνει ότι το επιπρόσθετο διοικητικό κόστος και άχθος για τις εταιρείε ελαχιστοποιείται, γιατί προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουλέψουμε πάνω στις συστάσεις της έκθεσης ΠΕΠΣ e του ΩΣΑ, το οποίο σημαίνει ότι το ίδιο πρότυπο, ε, το ίδιο στάνταρ, ο ίδιος κανόνες ε, εφαρμόζονται όχι μόνο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα λοιπά μέλη του ΩΣΑ. Και αυτό μειώνει το διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις, γιατί εναρμονίζονται τα προαπαιτούμενα κείμενα ή προϋποθέσεις σε σχέση με την ανταλλαγή των στοιχείων, ποια στοιχεία πρέπει να ανταλλαχθούν και με ποια μορφή πρέπει αυτά να υποβληθούν. Και η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βεβαίως είναι να μειώσει το διοικητικό βάρος όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τηρείται η αρχή της επικουρικότητας γιατί σαφέστατα το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να επιληθεί σε επίπεδο ενός μόνο κράτους μέλους, χωρίς συνεργασία μέσα στην ε, ίδια ομάδα χωρών, η αποτελεσματικότητα είναι πολύ αμφισβητούμενη χωρίς τη συνεργασία περισσότερων χωρών. Τώρα, σε γενικές γραμμές ως εισηγητής βεβαίως και στηρίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να προτείνω δύο ε, ίσονος σημασίας αλλαγές στο σχέδιο ε, κειμένου. Πρώτον, να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη διαδικασία και να είναι αποδέκτης αυτής της αυτόματης ανταλλαγής από χώρα σε χώρα. Δηλαδή, Σήμερα, οι πολυεθνικές που έχουν την έδρα τους σε ένα κράτος μέλους ε, είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν ε, ε, έκθεση με τις δραστηριότητες τους αναχώρα, τις δραστηριότητες των θυγατρικών τους ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών από τη στιγμή που η πολυεθνική έχει ιδιοκτησία μετοχικού κεφαλαίου σε κάποια άλλη εταιρεία. Επομένως, ε, πρέπει να υποβάλει όλα αυτά τα στοιχεία η πολυεθνική, η εταιρεία σε όλες τις χώρες, τις φορολογικές αρχές ε, των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται εγώ προτείνω πέραν των ε, φορολογικών αρχών να, είναι, να να τα υποβάλει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα στοιχεία, γιατί η Επιτροπή είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται αυτή η οδηγία. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει όλα τα στοιχεία διαθέσιμα για να μπορέσει να διασταυρώσει σε ποιο βαθμό γίνεται πράγματι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Και η δεύτερη πρόταση που υποβάλλουμε στην έκθεσή μας είναι ότι θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια μετά από ένα έτος εφαρμογής αυτής της οδηγίας να έρθει και να ε, κάνει αναφορά και στο Συμβούλιο αλλά και στο Κοινοβούλιο για το κατά πόσο τα μέτρα αυτά υπήρξαν αποτελεσματικά. Και ζητώ ως εισηγητής να υποβάλει έκθεση για την αποτελεσματικότητα αναχώρα, σε ποιο βαθμό πράγματι εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες μας και περιορίσαμε τελικά το εύρος των επιβλαβών φορολογικών πρακτικών των εταιριών μέσω του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τους σοσιαλιστές και ο ο κ. Μορέλ, κάποιος τέλο πάντων. Θέλετε το λόγο. Λίζα, ε, θα είμαι πολύ σύντομη. Πολύ καλά αυτά που είπε ο εισηγητής. Σύμφωνο με τις ανησυχίες και τις παρατηρήσεις σας για το ότι το Συμβούλιο προεξόφλησε τη θέση του Κοινοβουλίου, ενώ το Κοινοβούλιο ήταν ε, βασικός δρόν στην ε, πρόθεση της λογοδοσίας της διαφάνειας και ενός νέου πολιτικού πλαισίου σε θέματα άμεσης φορολογίας που σχετίζονται άμεσα με αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό η πρωτοβουλία αυτή να συνδέεται με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε αναλάβει σε φορολογικά ζητήματα, όχι μόνο στην Επιτροπή Τάξε, αλλά και στα διαδοχικά νομικά κείμενα που θα εξετάσει η ΕΚΟΝ. Τούτο προκύπτει από την... και που προκύπτουν από την πολιτική πίεση και τα ευρήματα της τάξε 1 καθώς και από την διαδικασία που ακολουθούμε στην τάξε 2. Ζητούμε λοιπόν να υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση της Επιτροπής αυτής στην διαδικασία που ακολουθείται στο Κοινοβούλιο. Πιο συγκεκριμένα, για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα, θέλω να καλωσορίσω μία από τις προτάσεις του εισήγητη να εμπλακεί η Επιτροπή πολύ περισσότερο στη διαδικασία αυτή. Είναι σημαντικό κατόπιν να παρακολουθούμε την έκθεση χώρας προς χώρα για τις υπερεθνικές. Χτες είχαμε κάποιους σημαντικούς εμπλεκόμενους ε, ε, που μίλησαν για το θέμα αυτό στην Επιτροπή 2. Η λογοδοσία και η αναχώρα έκθεση πρέπει να δημοσιοποιείται αυτό είναι το βασικό στοιχείο της επιχείρησης. Η διαφάνεια λοιπόν πρέπει να γίνεται κατανοητή από τις πολυεθνικές και από τους πολίτες και τις φορολογικές αρχές. Η διαδικασία είναι μόνο μία αφετηρία αυτή, ξεκίνησε καλά, αλλά πρέπει να ακολουθηθεί από σειρά εξελίξεων που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και δημιουργούν νέα φιλοσοφία, νέα ατζέντα, νέα πρακτική σε ό,τι αφορά την άμεση φορολογία και τον συνδυασμό μεταξύ μεγαλύτερης ενοποίησης και ταυτόχρονα σεβασμού της ομοφωνίας που, που απαιτείται στα θέματα άμεσης φορολογίας. Σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου πρέπει να γίνεται σεβαστός και να ενισχύεται. Ταυτόχρονα ως Κοινοβούλιο ήμασταν σαφείς στην ανάγκη να υπάρχουν συγκλίνοντα μηνύματα και συνοχή των κειμένων που υιοθετούμε απαντώντας Στι πρωτοβουλίε τη Επιτροπή και τι αποφάσεις του Συμβουλίου. Αυτό είναι ο λόγο που είναι σημαντική η αρχική παρατηρήση του Πρόεδρου. Ευχαριστώ. Υπήρκο Ρούχονεν Λέρνερ. Πρόεδρε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το κείμενό του. Οι τροπολογίε του κ. Ροζάτη ιδίω διατηρούν την ισορροπία που είχε προσπαθήσει να προωθήσει η Επιτροπή στο αρχικό της κείμενο για τις αναχώρα εκθέσεις. Η πρόταση του εισηγητή να συμπεριληφθεί η Επιτροπή ως μέρος του, με, της ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει να υποστηριχθεί. Δεν αλλάζει τα καθήκοντα της Επιτροπής. Τα κράτη είναι αυτά που έχουν τη βασική ευθύνη. Εγώ εκπροσωπώ το ίσια, εδώ έχουμε διαφορετικές απόψεις ωστόσο. Σύμφωνα με την ομάδα η αιτήσια έκθεση της Επιτροπής ήταν αρκετή. Η Ένωση πρέπει να ακολουθήσει τη δουλειά που κάνει ο ΣΑ στον τομέα της φορολογίας, ιδίως ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, τα κράτη-μέλη του ΟΣΑ εφαρμόζουν τις συστάσεις BEPS. Και το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και έκθεση αναχώρα. Εγώ προσωπικά ωστόσο υποστηρίζω την δημοσιοποίηση των εκθέσεων αναχώρα για την φορολογία. Ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα είναι βάση για να αποφύγουμε την ε, μεταφορά των ε, κερδών και την διάβρωση της φορολογικής βάσης. Η Ένωση έχει περιορισμένη αρμοδιότητα στα φορολογικά ζητήματα αλλά είναι κρίμα που το Συμβούλιο δεν ακούει επαρκώς το Κοινοβούλιο στον τομέα αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για το πρόβλημα αυτό. Thank you for the ALDE group, για την Άλντε, η κόρα. Και εγώ ξεκινώ συγχαίροντας τον εισηγητή. Εξαιρετική δουλειά έκανε ο κ. Ζουζάτη. Τα αποτελέσματα είναι γρήγορα. Παρότι είμαι ε, υποστηρίζω να στείλουμε επιστολή στον κύριο Ντάιζεμπλουμ που είναι πάντα χαρούμενος όταν προχωράει γρήγορα το Συμβούλιο, αλλά να του πούμε ότι ε, ότι πρέπει να περιμένει και εμάς Δεν, ε, η ταχύτητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να γνώμε το Κοινοβούλιο. Υποστηρίζουμε τις συστάσεις BEPS. Τα σημαντικότερα λόγια στην οδηγία, στην οδηγία αυτή είναι οι λέξεις υποχρεωτική και οι λέξεις αυτόματη. Πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα επίσης η έκθεση να μας παρουσιάζει ένα απολογισμό όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα αλλά και το πώς δουλεύει. Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε το διοικητικό βάρος. Ταυτόχρονα με ενδιαφέρουν επίσης ε, και το πόσο αποτελεσματικά είναι όλα αυτά. Η ανταλλαγή τώρα γίνεται τώρα γίνεται υποχρεωτική και αυτόματη. Θα ήθελα να δω τι συνέπειες θα έχει αυτό, γιατί ακούμε κατηγορίες να αλληλοκατηγορίες μεταξύ των κρατών. Θα ήθελα να ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτή τη αυτόματης ανταλλαγή στοιχείων. Πάντω υποστηρίζουμε πλήρω την έκθεση Ροζάτη. Ευχαριστώ. Ο Μιγγέλ Μπιέγκας για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Μιλάμε για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν είναι πρόσφατο το θέμα. Ήταν αντικείμενο της οδηγίας για, του, 2003 για την ε, οι ε, οδηγίε για την επαγγελματική απασχόληση του 2012, τον συνεργατών του ΩΣΑ. Ε, συζητάμε τα θέματα αυτά από τη δεκαετία του 80, τότε πρωτοβγήκαν οι πρώτες προτάσεις. Δεν είναι κάτι νέο λοιπόν. Γιατί όμως μέχρι τώρα δεν εφαρμόστηκε τίποτα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα νομίζω που πρέπει να θέσουμε. Κατά την άποψή μου, η ομάδα εργασίας του ΕΚΟΦΗΝ ε, στην ε, συνάντηση ε, που ήταν και κλεισμένο το φινογείο του ΕΚΟΦΗΝ αναφέρθηκε ότι 26 χώρε δεν είχαν ποτέ κάνει μια τέτοια δήλωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το νομοθετικό πακέτο δηλαδή είναι χρήσιμο, πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Η ενημέρωση πρέπει να είναι δημοσιοποιημένη διότι εμείς πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα η κοινή γνώμη είναι αυτή που είναι κινητήρια δύναμη των μεταρρυθμίσεων που ε, χτυπούν την ε, φοροδιαφυγή. Το ανώτατο όριο είναι επίσης πολύ ψηλό, αφήνει εκτός μεγάλο μέρος των πολυεθνικών το ανώτατο όριο πρέπει να μειωθεί για να καλύψει περισσότερες επιχειρήσεις. Συνολικά, πιστεύουμε ότι είναι ένα θετικό βήμα, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερο για να μην επαναληφθούν το παρελθόν για τους πράσινους. Πρόεδρε, Συγχαρητήρια προς τον κύριο Ροζάτη. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κόρα. Μας απογοητεύει ο τρόπος που το Συμβούλιο πέτυχε πολιτική συμφωνία. Αλλά το ότι μας αγνόησε νομίζω ότι είναι κάπως εξευτελιστικό. Ευχαριστώ τον εισηγητή που ετοιμάζει ένα σχετικό κείμενο. Τρεις ανησυχίες έχουμε με την έκθεση. Πρώτον, εμβέλεια της οδηγίας. Ο ορισμός των μεγα... τον ορισμό των μεγάλων επιχειρήσεων, τις κυρώσεις και την εμπιστευτικότητα. Για την εμβέλεια, το πεδίο εφαρμογή. ίσως ε, οι σοσιαλιστές να μας υποστηρίξουν αυτό εμάς, μας ανησυχεί το ότι θα πρέπει τουλάχιστον να ακολουθήσουμε την οδηγία, τον ορισμό για τις μεγάλες επιχειρήσεις που βρίσκουμε στην οδηγία για τα λογιστικά πρότυπα. Επίσης, θα έπρεπε αυτό να επεκταθεί περαιτέρω. Τι σημαίνει μικρομεσαία επιχείρηση στο πλαίσιο αυτό της, ενημέ... της απέτησης φορολογικής ενημέρωσης. Μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αφέμητο φορολογικό επιζήμιο, φορολογικό ανταγωνισμό και ξέρουμε οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν νομίζω να είναι το ίδιο. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις δεν βλέπουμε ότι έχει σωστά μέτρα εφαρμογής επιτροπή που δεν μπορούν να προκύψουν αν δεν δώσουν ε, τα κράτη-μέλη και οι επιχειρήσεις της πληροφορίας, οι επιχειρήσεις της στα κράτη-μέλη. Εμείς θα προτείνουμε λοιπόν έναν, ε, μια μορφή παρακράτησης φόρου των χρηματοοικονομικών οργανισμών σε τρίτους χώρες που δεν παρέχουν ε, πληροφορίες, ε, ανταλλαγή πληροφοριών στην Ένωση που είναι ένα αντίστοιχο με μια διαδικασία στη ΣΥΠΑ που φορολογούν τις συναλλαγές που φεύγουν από τη ΣΥΠΑ αν δεν υπάρχει φορολόγηση, στοιχεία για τη φορολόγηση στη χώρα ε, άφηξης, την εμπιστευτικότητα. Δεν πρέπει αυτό να χρησιμοποιηθεί σαν πρόσχημα για να εμποδίσουμε την ε, διαφάνεια συνολικά. Η αναχώρα ενημέρωση δεν περιλαμβάνει εμπορικά μυστικά. Δεν μπορούν οι χώρες να χρησιμοποιήσουν αυτό ως επιχείρημα για να μην υποβάλουν εκθέσεις και θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες. Επίσης θα εξετάσουμε τροπολογίες για την δευτερογενή ενημέρωση για τις υποκατάστατες των ε, θηγατρικών και για τους πράσινους η αυτόματη ενταλλαγή πληροφοριών αναχώρα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, αλλά δεν είναι η πλήρης αξιολόγηση, ετήσια αξιολόγηση που θέλουμε να δούμε. Ευχαριστώ. Uh, Catch the Eye. Oh, sorry, sorry. First, uh, yes, is Kappel. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, auch ich begrüße die Initiative des Kappel. Καλή η πρωτοβουλία του εισηγητή να, στέλνει, να στείλει επιστολή στον κύριο Ντάισεμπλουμ. Δεν είναι αποδεκτό το Συμβούλιο να αγνοεί τα καθήκοντά του εδώ και να αποφασίζει πριν το δούμε εμείς. Η έκθεση είναι ισορροπημένη. Αντιμετωπίζει το θέμα των αιτήσεων ε, αξιολογήσεων και επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την επιθετική φορολογική, ε, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Είναι ένα από τα τέσσερα μέτρα για να αντιμετωπίσει η Επιτροπή την φοροαποφυγή και τις νέες μορφές φοροαποφυγή, φοροαποφυγής καθώς και την υλοποίηση της οδηγίας για τις ε, ε, μορφές αντιμετώπισης της φοροαποφυγής ακολουθώντας τις προτάσεις BEPS τα μέτρα που ανέφερα περιέχουν και πρόσθετα μέτρα. Τώρα για την έκθεση. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις, δηλαδή 750 εκατομμύρια κατόφλι στον συνολικό τζίρο της επιχείρησης, μου φαίνεται σωστό. Και σε ό,τι αφορά την φορολογική αρχή, δηλαδή την βασική αρχή της φορολόγησης. Αυτά μου φαίνεται ότι είναι σκόπιμα. Το ίδιο η έκταση της ανταλλαγής πληροφοριών, διότι δηλαδή όλα τα δεδομένα τα οποία έχουν σχέση με τον, με τον φόρο, με τη φορολογήση, ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να είναι κάπως πιο φιλόδοξο. Νομίζω ότι το 12 μήνο είναι υπερβολικά μακρός χρόνος. Χρειάζεται πολύ συντομότερος χρόνος για την υποβολή των σχετικών εκθέσεων και θα προτείνω λοιπόν η υποβολή των εκθέσεων αναχώρα να γίνεται ταυτόχρονα, στο τέλος δηλαδή του πρώτου τριμήνου, με την υποβολή των ισολογισμών. Ότι βασίζεται τώρα στις προτάσεις του ΟΣΑ μου φαίνεται σωστό. Μου αρέσει δε η πρόταση, δηλαδή πριν να ληφθεί απόφαση, να γίνεται υπολογισμός του κόστους. Θα πρέπει να γίνεται τον Απρίλιο αυτό, δηλαδή αμέσως μετά από το πρώτο τρίμηνο. Και αυτή την εκτίμηση να τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Γιατί αν το κόστος υπερβαίνει το όφελος, τότε είναι λάθος ο στόχος. Μια έκθεση τώρα, μια μάλλον πρόταση του εισηγητού που δεν επιθυμώ να υποστηρίξω, είναι η αυτόματη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, να μην υποβάλλονται εκθέσεις μονάχα στις αρμόδιες αρχές των χωρών, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συντάσει την βάση τους έκθεση. Δεν διακρίνω εδώ καμιά προστιθέμενη αξία. Είναι σημαντικό η Κομισιόν να αναφέρει σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου για την φοροαποφυγή και εν προκειμένου να, γίνονται, να ε, κατατίθεται και παραδείγματα. Είμαι όμως αντίθετη με την αυτόματη αυτή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Συγγνώμη Επιτροπής ε, ως παραλήπτρια των εκθέσεων αναχώρα. Σας ευχαριστώ. Μορέλ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη γιατί είχα ένα πρόβλημα στις συγκοινωνίες για να έρθω, γι' αυτό καθυστέρησα. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ροζάτη για το κείμενό του που επιτρέπει στις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν πρόσβαση στις δηλώσεις αναχώρα των εταιριών. Τον ευχαριστώ επίσης για την επιφυλακτικότητά του έναντι της δράσης του ε, Συμβουλίου. Φοβόμαστε ότι θα επαναληφθεί το σενάριο DAC 3 τα κράτη-μέλη δεν έχουν υιοθετήσει επισήμως τη συμφωνία, αλλά βρήκαν ένα τεχνικό συμβιβασμό χωρίς τη γνώμη του Κοινοβουλίου και είναι θέματα στα οποία ε, το Κοινοβούλιο ε, θέλει να αποφανθεί. Η πρόταση του Μοσκοβισή είναι μια καλή βάση, δείχνει ότι έχει ξεκινήσει μια σωστή δυναμική. Εμείς τι ξεκινήσαμε εμείς οι Ευρωπαίοι με την κινητοποίηση της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Τα πράγματα πηγαίνουν λοιπόν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, πιστεύω ότι μπορούν ακόμα να βελτιωθούν και θα ήθελα να σας παρουσιάσω δύο παραδείγματα. Πρώτον, έχουμε το reporting αναχώρα. Να είναι δημόσια τα δικαιώματα των μετόχων. Δεν είναι αυτό το αντικείμενο της οδηγίας που συζητούμε τώρα, Μιλούμε για την εδραίωση της διοικητικής συνεργασίας. Είναι όμως δικιά μας υποχρέωση να έχουμε μία δέσμη κειμένων συνεκτική, να υπάρχει συνοχή μεταξύ των περιεχομένων των διαφόρων νομοθετικών κειμένων. Και ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως είναι το εξής. Η διαφάνεια δεν μπορεί να αφορά μόνο το 10 και 15% των πολυεθνικών, παρόλο που αυτές έχουν το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. Η λειτουργία της ενιαίας αγοράς βασίζεται στην ίση μεταχείριση μεταξύ των εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις γίνεται. Γι' αυτό να πάρουμε το κατόφλι των επιχειρήσεων που προβλέπεται στην οδηγία ε, για τα δικαιώματα των μετόχων και τα λογιστικά, δηλαδή 250 απασχολούμενοι και κύκλος εργασιών 40 εκατομμύρια ευρώ. Και θα πρέπει οι προϋποθέσεις να είναι εξίσου ακριβείς με αυτές που ζητούμε για τα δικαιώματα των μετόχων και για το reporting αναχώρα. Και θα ήθελα να προσθεθούν και κάποιοι άλλοι δείκτες, όπως είναι οι ενισχύσεις ενδεχομένως που λαμβάνουν. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να πω ότι μία από τις αποστολές μας είναι να έχουμε ένα αποτελεσματικό ε, και παραγωγικό νομοπαρασκευαστικό έργο. Το DAC 4 είναι γεμάτο εξαιρέσεις και απαλλαγές κάθε είδους. Τα κράτη-μέλη θέλουν να διατηρήσουν και τη δυνατότητα το ένα κράτος να αρνείται την, κατα... την πληροφορία στο άλλο κράτος μέλος και αντίστροφα. Όλα αυτά είναι μηχανισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το FACTA. Εγώ πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη ε, ήδη έχουν ξεκινήσει να λένε ότι το reporting είναι δευτερεύον. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Αυτά με δύο λόγια. Σε κάθε περίπτωση Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε εικονοποιημένοι με την δράση μας. Αναφεσβήτητα τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λογική και σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριο Στρεμόζα. Okay, so Mr. Sí. Gracias, Presidente. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου. Πιστεύω ότι πράγματι το Συμβούλιο δεν διανοείται την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παρακολούθηση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών και θεωρώ ότι αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό για τρεις λόγους. Καταρχάς, τα στοιχεία αυτά δεν αντιστοιχούν με την ενιαία αγορά. Δηλαδή, δεν θα δώσουν τα κράτη-μέλη πληροφορίες για τη δική τους φορολογική πολιτική, για τη φορολογική πολιτική που ακολουθεί το κάθε κράτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προστατεύσει τις συνθήκες της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Αυτό καταρχάς είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Δεύτερο, πολλές από αυτές τις πολιτικές έχουν σχέση με αυτό το οποίο ονομάζουμε κρατικές ανισχύσεις. Και υπ' αυτή την έννοια ο αρμόδιος επίτροπος είναι αυτός που πρέπει αυτά να τα εξετάζει προσεκτικά και να δει κατά πόσο τα tax rulings, οι ειδικές φορολογικές συμφωνίες μεταξύ κράτους και χι επιχείρησης αποτελούν ένα είδος κρατικής ενίσχυσης. Ε, και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύσει το ρόλο της να έχουμε μία ε, ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, έστω και σε εμβριακή μορφή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Η Επιτροπή θα πρέπει να ε, το διαρθρώσει αυτό στα αρχικά του στάδια. Στη διακυβέρνηση του ευρώ όλα συντείνουν έτσι ώστε να έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Το να στερήσουμε ε, ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ρόλο του συντονισμού είναι κάτι που αντιβαίνει στο ρου της ιστορίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος γιατί τα βασικά έχουν ήδη υποθεί ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσωπώ πολίτες πολύ συνειδητοποιημένους θέλω να επισημάνω το εξής. Συμφωνώ απολύτως με τα λεγόμενα του Σκιώδη εισηγητή, με τη φίλη Κόρα και με τους λοιπούς. Ωστόσο, το θέμα αυτό δεν είναι μόνο τεχνικό. Πολύ καλά έχουν κάνει τη δουλειά τους όλοι οι σκιώδεις εισηγητές, ο εισηγητής και τα λοιπά σε τεχνικό επίπεδο. Όμως το θέμα είναι ξεκάθαρα πολιτικό και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Ροζάτη να μην το ξεχνάει και οι υπόλοιποι να μην το ξεχνούν. Σήμερα η Ευρώπη χάνει έδαφος και πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να ελπίζει κανείς και να επιθυμεί πραγματικά να είναι πολίτης της ευρωπαϊκής οικογένειας. Να εμπνεύσουμε αυτό το όραμα μιας Ευρώπης πιο ενοποιημένης, πιο ολοκληρωμένης, πιο ενιαίας. Και με αυτό τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Εάν δεν παρέμβουμε, ενδεχομένως, Εάν η Κομισιόν δεν παρέμβει ενδεχομένως σε αυτό το τομέα είναι κάτι το πολιτικός απαράδεκτο. Αποτελεί πρόκληση από το Συμβούλιο το οποίο τελικά ε, μεταστρέφεται και γίνεται εχθρός της άποψης που θέλει περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Ε, καθαρά πολιτικό του ζήτημα και έχει τεράστια πολιτική σημασία. Ευχαριστώ, ο Πέτερ Ζήμων, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με ορισμένους από τους, συμφων... τους ε, Η διαφάνεια είναι πολύ σημαντικό, αλλά η διαφάνεια έχει νόημα όταν και η αρχή η οποία θα συναγάγει τα συμπεράσματα από τη διαφάνεια συμμετέχει και αυτήν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν η αυτόματη κατάθεση των ε, εκθέσεων δεν περιλαμβάνει αυτομάτως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε οι γκρίζες αυτές ζώνες θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και οι χώρες μέλη οι οποίες φρόντισαν στο παρελθόν να στερήσουν φορολογικά έσοδα από άλλες χώρες μέλη θα συνεχίσουν να ζουν και να βασιλεύουν. Αν θέλουμε ε, διαφάνεια, αν θέλουμε tax ruling, που αν θέλουμε να πάψουν μάλλον τα tax ruling, τότε πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η μόνη η οποία διαθέτει και το ξύφος από τις συνθήκες για να επιβάλλει τον νόμο, θα πρέπει να είναι και αυτή αυτομάτως το σύστημα. Οι χώρες που δεν το υποστηρίζουν αυτό, ή επίτηδες δεν θέλουν, ή τελικώς συμπαρασύρονται και συμπορεύονται με τους άλλους. Ευχαριστώ πολύ. Τρεμόζα. Έχετε ζητήσει για αυτό το, συζήτηση για το θέμα αυτό, όχι. Τώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί την Επιτροπή Οικονομικών και τον κύριο Ρωσάτη ιδιαίτερα για το έργο σας. Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της διαφάνειας είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία στη στρατηγική της Κομισιόν για την καταπολέμηση της, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Ε, το εργαλείο που προβλέπεται στην έκθεση είναι σημαντικό με στη στρατηγική αυτή. ΤΑΚ 2 και ΤΑΚ 3, και, όπως τα είπατε, και ΤΑΚ 4 τώρα, είναι σημαντικά βήματα που έγιναν για να προσφερθούν, να παρασχεθούν μάλλον οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες στις φορολογικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εκτιμά ιδιαίτερα την ε, επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους τομείς αυτούς και ελπίζει ότι αυτό θα συνεχιστεί και για τα επόμενα νομοθετικά βήματα. Βεβαίω και χρειάζεται ταχεία πρόοδος. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό είναι πολύ θετικό. Το ειδικό αυτό θέμα, για το SWIFT δηλαδή, έχει συζητηθεί ήδη από καιρό και στον ΩΣΑ και μεταξύ άλλων δικαιοδοσιών. 20 από 28 χώρες μέλη έχουν ήδη συνυπογράψει την ανταλλαγή αυτή πληροφοριών. Οι περισσότερες από αυτές διαθέτουν ήδη εθνική νομοθεσία ή την εξελίσσουν. Θα προχωρήσει λοιπόν, θεωρεί η πρόοδος αυτή, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά βέβαια ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για την ουσία. Είπατε κι εσεί ότι η δεσμευτική ανταλλαγή πληροφοριών είναι πολύ σημαντική. Και οι πληροφορίε που ε, παρέχουν οι φορολογούμενοι στις φορολογικές αρχές, αλλά και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών. Το κείμενο είναι σωστό από την άποψη αυτή ακούστηκαν και άλλα σχετικά με το ουσιώδες περιεχόμενο της προτάσεως. Θα μιλήσω για τρία. Η πρόταση της Επιτροπής βασίστηκε στην σύσταση που συμφωνήθηκε στον ΟΟΣΑ, ε, Action 13. Υποστηρίζουμε το κείμενο που συζητήθηκε στον οργανισμό αυτό με καθαρό στόχο να μην δημιουργηθεί ένα πρόσθετο στρώμα για υποβολή εκθέσεων αναχώρα από τις πολυεθνικές. Αλλά κατέστη σαφές με την πρόταση ότι οι ευρωπαϊκές αλλά και μη ευρωπαϊκές πολυεθνικές οι οποίες ωστόσο δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά θα πρέπει να παίζουν με τους ίδιους κανόνες. Και αυτό διαφυλάσσεται και στο συμβαστικό κείμενο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το πεδίο εφαρμογή, το περιεχόμενο των πληροφοριών, την περιοδικότητα των ε, συναλλαγών, το ΤΑΚ 4 συμμορφούνται με τις ε, συστάσεις του ΩΣΑ και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για μας. Δεύτερο, ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη ορίζεται στην DAC Directive Administrative Cooperation και στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να παρακολουθεί την λειτουργία της οδηγίας αφού υποχρεώνονται οι χώρες μέλη σε αιτήσια βάση να παρέχουν πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά ενδεχόμενα κολλήματα τομείς που χρήζουν βελτιώσεως και αυτά θα τα αναλύει σε τακτική βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπροσθέτως στις DAC 4 η Κομισιόν θα λαμβάνει πληροφορίες από τις χώρες μέλη και για πολυεθνικούς ομίλους που αρνούνται να υποβάλουν σχετικές πληροφορίες. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, πιστεύουμε εμείς, για να διασφαλιστεί ώστε η ε, ανταλλαγή πληροφοριών θα λαμβάνει χώρα πράγματι στην πράξη. Τρίτο, το εάν Τώρα, πρόσθετες οργανώσεις ε, ενδιαφερόμενων μερών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ε, στις προφορίες αυτές είναι ξεχωριστό ερώτημα και βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό επεξεργασία στον αγωγό καθώς λέμε και έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει την εργασία που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελέτη αντικτύπου στην νομική πρόταση για το δημόσιο CBCR. Όταν θα εγκριθεί λοιπόν αυτό, ένας αριθμός όλοι δηλαδή στην ουσία ενδιαφερόμενοι θα, stakeholder δηλαδή, θα έχουν πρόσβαση πληροφορίες αυτές. Και αυτό απαντά έτσι στην ερώτηση αν δηλαδή η Κομισιόν θα πρέπει να προχωρήσει στην ε, υποβολή αναφορών αναχώρα. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι, ευχαριστώ για την έκθεση του Κοινοβουλίου και αναμένουμε την συνέχιση της επικοδομικής αυτής συνεργασίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επιτροπή. Κύριε Σιγητά τελευταίες σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ πρώτα όλους τους παρεμβάντες, ιδίως δε τις, ε, ε τους ηγητές για τα επικοδομητικά του σχόλια. Βλέπω να διαγράφεται ευρεία υποστήριξη για το μέτρο, για το μέτρο αυτό DAC 4. Αυξάνεται η κατανόηση ότι δεν μπορούμε να αγωνιστούμε αποτελεσματικά κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τακτικές και πρακτικές φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, αν δεν έχουμε αναχώρα υποβολή εκθέσεων προς τις φορολογικές αρχές, αλλά και να έχουμε και ένα μηχανισμό για την ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών μεταξύ χωρών μελών. Είναι λοιπόν σημαντικό συμπέρασμα αυτό, ότι, χρειάζεται, ότι υπάρχει μάλλον ευρεία ε, στήριξη αυτού του μέτρου. Ευχαριστώ όλες και όλους που υποστήριξαν την πρωτοβουλία μας για να εκφράσουμε δηλαδή δυσαρέσκεια απέναντι στην κίνηση του Συμβουλίου να βάλει την πολιτική απόφαση πριν από τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό όχι μόνο για λόγους διαδικαστικούς αλλά, αλλά και όπως είπε και ένας εκ των ομιλητών για να εξασφαλίσουμε συνοχή και συνεκτικότητα του έργου μας σε όλο το φορολογικό πακέτο. Ένα άλλο θέμα που ίσως συγκεντρώνει λιγότερη συνένεση, αλλά θα συζητηθεί πάντως στη διάρκεια των εργασιών μας με τους και Ένα θέμα είναι η πρόσβαση, η δημόσια πρόσβαση στις προφορίες αυτές. Αναμένουμε ακόμα την μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ελέγχθη και προτείνω το θέμα αυτό να αναμείνει η συζήτηση σε ευθετότερο χρόνο. Οι περισσότεροι εκ των ομιλητών στήριξαν την ιδέα ότι μέρος της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν και ορισμένες φωνές που προτείνουν το αντίθετο. Η μόνη δικαιολογία για να είναι μέρος της διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι δηλαδή πραγματικός στα χέρια της ο μηχανισμός να ελέγχει την λειτουργία της οδηγίας και σε ποιο βαθμό εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους οι χώρες μέλη σε ό,τι αφορά τις ανταλλαγές των πληροφοριών από την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μείνει εκτός της διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, είμαι ανοιχτός σε συζήτηση. για ορισμένα από τα άλλα θέματα τώρα. Το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Επίσης τέθηκε σε συζήτηση για πιο σε ποιο βαθμό μάλλον το προτινόμενο κατόφλιο των 750 εκατομμυρίων κύκλου εργασιών αρκεί για να καλύψει όλες τις πολυεθνικές. Κάποιοι ή κάποιες είπαν να μειωθεί το κατόφλιο. Ίσως, αλλά το βασικό επιχείρημα υπέρ τούτου δότου ποσού είναι για να είμαστε σύμφωνοι με τις ε, οδηγίες BEPS του ε, ΟΣΑ για να μην επιβαρύνουμε επιπρόσθετα ή να βάλουμε κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μειονεκτική θέση απέναντι σε μη ευρωπαϊκές πολυεθνικές. Είναι καλύτερα να υπάρχει ένα στάνταρτ κατόφλιο που να εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις και αυτές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων που είναι εκτός. Αυτή είναι η εξήγηση που έχω να σας δώσω. Για τις κυρώσεις ένα ενδιαφέρον θέμα είναι σε ποιο βαθμό είμαστε διατεθειμένοι να ελέγξουμε και να επιβάλλουμε την εφαρμογή της οδηγίας. Θέμα το οποίο μπορεί να συζητηθεί κι άλλο. Ε, μια ενδιαφέρουσα πρόταση έγινε επίσης για την περίπτωση παρακράτησης χώρων και μπορούμε εκεί να το ξανασυζητήσουμε. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα, να υπενθυμίσω ότι η οδηγία υποτίθεται ότι θα μεταφερθεί σε εθνικές νομοθεσίες μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους. Αυτό συμβαίνει ταχεία διαδικασία. Υπάρχει και η πρόταση για την υποβολή των αναχώρα εκθέσεων στις ε, φορολογικές αρχές είναι ένας χρόνος μετά από το οικονομικό έτος. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι σωστή η ε, ρύθμιση αυτή. Άλλωστε μας δεσμεύουν οι προτάσεις BEPS του ΩΣΑ που περιλαμβάνουν το 12 μήνο. Και πάλι όμως δεν θέλουμε να βάλουμε δύο πρότυπα, δύο στάνταρτ και να χωρίσουμε έτσι τις επιχειρήσεις σε δύο ομάδες έγιναν και άλλα σχόλια τα οποία εξετίμησα ιδιαίτερος. Δεν έχω έτοιμες απαντήσεις για όλα τα θέματα που θέσατε. Χαίρομαι όμως που ε, διαμορφώνεται μια γενική ε, συνένεση σε ό,τι αφορά την ανάγκη της νομοθετικής ρύθμισης και αναμένω την περαιτέρω συνεργασία με τους ε, συναδέλφους Σκιώδης Ισηγητάς ε, με την ελπίδα ότι το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής θα είναι θετικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρονοδιάγραμμα ως εξής. 21η Τρίτου στις 5 το απόγευμα κατάθεση τροπολογιών. 25 Απριλίου συζήτηση. 26 στην, ε, στην συζήτηση Επιτροπή και ψήφος την 1η Μαΐου. Θέμα 5 της ημερήσιας διάταξης τώρα έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ετήσια έκθεση 2014. Η συγκεκριτής είναι ο κύριος Τρεμόσα. Έχετε το λόγο αγαπητέ κύριε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, ήταν χαρά μου να ετοιμάσω το σχέδιο γνωμοδότησης και ελπίζω να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας για το θέμα αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 4.000 καταγγελίες για πιθανή παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ε, οι περισσότερες αφορούσαν την Ισπανία, 500, και από πίσω η Ιταλία. Από το 2013 και μετά άνοιξαν περίπου 3.000 διαδικασίες παραπομπής ε, από την Επιτροπή λόγω παραβίαση 439 οδηγιών. Οκτώ κράτη-μέλη στην πραγματικότητα ε, κατά μέσο όρο παραβιάζουν τις, ε, μια οδηγία μετά το Μάστριχτ. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε συνάδελφοι είναι το εξή: Είναι τόσο μη αποτελεσματικό το, η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχουμε τόσο δυσκολία να υλοποιήσουμε αυτά που με τόσο δυσκολία εγκρίνουμε τα τελευταία χρόνια. Η πραγματικότητα είναι ότι στη, στον τομέα της οικονομίας και των χρηματοοικονομικών μόνο η Γερμανία σέβεται όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Αυστρία παραβιάζει μία οδηγία. Η κατάσταση για τις υπόλοιπες χώρες ωστόσο είναι κοντά στην, στη δραματική. 10 η Πολωνία, 9 το Λουξεμβούργο, 8 η Σλοβενία, 7 η Ισπανία κτλ. Το 2014 επιπλέον μόνο 10 από τις 157 βασικές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εφαρμόστηκαν πλήρως ή έδειξαν ουσιαστική πρόοδο. 6% δηλαδή ε, συντελεστή επιτυχίας. Επίσης υπάρχουν κράτη όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία που ακολουθούν περισσότερο τις συστάσεις του ΩΣΑ παρά τις συστάσεις κομισιών. Σας υπενθυμίζω ότι όσα είναι ένα think tank μόνο. Γι' αυτό το λόγο με την έκθεση ζητώ να ε, σταματήσει αυτό το τζαμπατζίδικο νομοθετικό καθεστώς όταν ένα κράτο παραβιάζει συστηματικά την ευρωπαϊκή νομοθεσία χωρίς επιπτώσεις. Ζητώ από την Επιτροπή να αντιδράσει για να επιβάλλει την νομοθεσία στα κράτη-μέλη και να μην θεωρούν τα κράτη ότι μπορούν να επιλέξουν τι τους αρέσει και τι όχι. Συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια δουλέψαμε σκληρά για να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση και τους σχετικούς κανόνες. Αν όμως η Επιτροπή δεν τολμά να χρησιμοποιήσει την δύναμη που έχει όταν κράτη-μέλη όπως η Γαλλία ή η Ισπανία δεν σέβονται τους δημοσιονομικούς στόχους, τότε τι κάναμε. Γιατί παράγουμε όλο ένα και περισσότερες οδηγίες όταν οι ήδη εγκριφίσεις παραβιάζονται συστηματικά. Στο, πρόγραμμα, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καταθέσεων ε, μπορούμε να προχωρήσουμε όταν 10 κράτη-μέλη αρνούνται να συμμορφωθούν με την υφιστάμενη νομοθεσία. Στο, στην νομοθεσία για την, ε, λύση των, για την ε, λύση των τραπεζών η οδηγία, η, τα κράτη-μέλη δεν σέβονται την οδηγία που θεσμοθετεί τα bail-in, ενώ η Ιταλία στην πρώτη ευκαιρία δεν την εφαρμόζει. Καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες γίνονται όλο και πιο ευρωσκεπτικιστές όταν στην, σε χώρες όπως η Ισπανία οι νομοθετικές ρυθμίσεις για, την, ε, για τις τράπεζες παραβιάζονται από όλες τις, από την κεντρική και τις περιφερειακές κυβέρνησεις. Σύμφωνα με την ε, Ισπανική Ένωση κατά τον ε, ε, καθυστερούμενων πληρωμών ε, χάθηκαν πάρα πολλές θέσεις εργασίας εξαιτία της μη συμμόρφωσης του κράτους με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν δεν εφαρμόζουμε την νομοθεσία, εφαρμόζουμε, μετατρέπουμε την Ένωση σε ένα τεράστιο think tank και οδηγούμε σε ε, πλήρη απο, ε, απονομιμοποίηση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Χρειαζόμαστε ισχυρότερες κυρώσεις κατά των κρατών μελών που δεν σέβονται την νομοθεσία, ιδίω στον τομέα των τραπεζών. Χρειαζόμαστε ουσιαστικού ελέγχου εφαρμογή ε, τη νομοθεσία από τι ίδιε κυβερνήσει, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί δρόντε για το μέλλον τη Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε μια νομοθεσία η οποία θα αντικατοπτρίζει τον δημοσιονομικό έλεγχο ε, σε οποιαδήποτε επιτροπή η συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας της Ένωσης ωστόσο πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά. Για την Επιτροπή νομίζω ότι ήρθε, τελείωσε η περίοδος της τεχνοκρατικής ε, προσέγγισης. Μπορούμε να ενισχύσουμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση της Ένωσης ε, αλλά αν δεν υπάρχει έλεγχος της εφαρμογής των νόμων όλα αυτά είναι μάτι. Ευχαριστώ για την ε, προσοχή σας. Περιμένω τα σχόλιά σας. Thank you very much. Actually, uh, parliamentary election normally can give strong legitimacy. Νομίζω ότι η κοινοβουλευτική εκλογή δίνει νομιμοποίηση, αλλά τέλος πάντων ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Για το ΕΛΚ. Κύριος Ζάκ. ευχαριστώ πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματο του κυρίου Ματουτσέλου που είναι ο Σκιώδης για το ΕΛΚΑ. Θα διαβάσω αυτά που σας προτείνει. Καλωσορίζουμε την γνωμοδότηση του κύριου Τρεμόσα ως εξαιρετική βάση για περαιτέρω δουλειά. Η σωστή υλοποίηση των, ε, της υφιστάμενης νομοθεσίας είναι κλειδί και συμφωνούμε με τον εισηγητή για τα ζητήματα που αναφέρει σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Δεν συμφωνούμε με την αναφορά όμως σε συγκεκριμένες χώρες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριος για τους σοσιαλιστές. Συνάδελφοι, ευχαριστώ τον εισηγητή για τη γνωμοδότησή του. Πολλές παράμετροι της γνωμοδότησης Τρεμόζα μας βρίσκουν σύμφωνος. Η εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης είναι βασική προϋπόθεση για να έχουμε μια ισχυρή Ένωση. Συμφωνούμε με αυτό. Το λένε και οι συνθήκες άλλωστε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα εκ νέου να υπογραμμίσω ότι και ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης έχει την ίδια νομική αξία με τις συνθήκες. Ωστόσο υπάρχουν κάποια σημεία όπου θέλουμε να προτείνουμε αλλαγές. Στην παράγραφο 3 υπογραμμίζω ότι η έλλειψη εφαρμογής ε, της οδηγίας για τις καθυστερούμενες πληρωμές ιδίως σε 11 κράτη-μέλη σχετίζεται και με την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών που επηρεάζονται από την κρίση. Ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στην εθνική νομοθεσία. Είναι σημαντικό η οδηγία για την πρόσβαση δραστηριότητε των πιστοτικών ιδρυμάτων και η προληπτική υποπτία τους η οδηγία για τις απαιτήσει δημοσιονομικού πλαισίου των κρατών μελών και η οδηγία για το δικαίωμα των καταναλωτών δεν έχουν υλοποιηθεί, δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα. Επιπλέον, στην παράγραφο 4, η ατελής φύση της Ευρωζώνης και της Ένωση είναι αυτή που δημιούργησε την κρίση στην Ένωση και η υπερβολική έμφαση σε μια συγκεκριμένη μορφή πολιτικής. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε, το Ευρω... διαμόρφωσε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την Τραπεζική Εποπτεία. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα έπρεπε να εφαρμόζεται καλύτερα, ιδίως από την χρήση της ευελιξίας και της ευκαμψίας. Βεβαίως δεν έχει ολοκληρωθεί η δουλειά. Χρειαζόμαστε πλήρη νομισματική ένωση, ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης συμφωνούμε ότι είναι σημαντική η τραπεζική κανονισμοί και σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας να εισάγετε μια ευρωπαϊκή διάσταση στο πρόγραμμα εγγύησεων των καταθέσεων, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εγγύησεων των Καταθέσεων. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να έχετε σε αντίφαση με την τραπεζική εποπτεία. Επιπλέον, η Υποστηρίζουμε την πρόσβαση της Επιτροπής στα στοιχεία για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Να συγχαρώ εκ νέου τον εισηγητή, προσβλέπω στην συνέχιση της συνεργασίας μαζί του και με τους άλλους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Um, uh, ευχαριστώ. Η συνάδελφος Κέι δεν μπόρεσε να είναι εδώ παρούσα. Μου ζήτησε να διαβάσω κι εγώ τα δικά της. τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Συμφωνεί ότι η αναφορά συγκεκριμένων περιπτώσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δεν εφαρμόζονται από κράτη-μέλη έχει τεράστια σημασία, το είπατε και εισαγωγικά. Αναφέρει ότι αυτό που ήταν εντυπωσιακό ήταν και ότι η και της συνεργασίας του ΜΥΦΙΔ 2 διαπίστωσε ότι τα κράτη δεν είχαν υλοποιήσει, δεν είχαν ενσωματώσει την ΜΥΦΙΔ 1. Ωστόσο, κατανοεί την καθυστέρηση κάποιων κρατών μελών στην εφαρμογή οδηγιών όταν θέτουμε υπερβολικά ταχείες ε, προθεσμίες είχε πάει σε μια συνάντηση γλωσσομαθών νομικών για την, τον κανονισμό για τα benchmarks, όπου ήδη το Συμβούλιο είπε ότι οι προθεσμίες ήταν υπερβολικά φιλόδοξες. Συχνά μιλάμε για better regulation, αλλά το είχε πει ο υπουργό, ο εκπρόσωπο του Συμβουλίου των Υπουργών, ότι θα βρουν ένα τρόπο να το προχωρήσουν γρηγορότερα, που δεν είναι μια σωστή προσέγγιση στα πλαίσια τη ε, Better Regulation. Προτείνει να υπάρξει ένα μεγαλύτερο όρο για το ΕΣΑΣ, ούτω ώστε να μπορεί να παρέχει περισσότερε πληροφορίε ε, στην Επιτροπή όταν έχει κάνει peer reviews για την εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης ε, στα διάφορα κράτη-μέλη και βρήκαν κενά στην υλοποίηση τον, ε, και εφαρμογή της νομοθεσίας. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που θέλει να κάνει. Τελευταία πρόταση στην έκθεση, για την έκθεση του εισηγητή είναι, ε, που θέλει να τονίσει και είναι ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει μια υποεπιτροπή της ΑΦΚΟ που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ίσως αυτό πρέπει να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο βέβαια. Γιατί τα θέματα αυτά εμφανίζονται αρκετές, ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν είμαι βέβαιος πώς ε, θα μπορούσε να παρακολουθήσει τόσο προσεκτικά μια υποεπιτροπή ένα τόσο εκτεταμένο θέμα. Ίσως να καταλήξουμε με στο τέλος να κάνουμε επικαλύψεις δραστηριοτήτων και όχι να το βελτιώσουμε. Ίσως ένας καλύτερος τρόπος θα ήταν να δουλέψουμε προς ε, ένα σύστημα που θα ζητούμε την Επιτροπή να ενημερώνει την ECOM τακτικά ή την οποιαδήποτε αρμόδια Επιτροπή για, για συγκεκριμένα θέματα και να παράσχουμε αυτό που αυτό στο οποίο στοχεύουμε δημιουργώντας ένα δημόσιο πλαίσιο συζήτησης και πώς βλέπει βέβαια να συνεργαστεί με τον εισηγητή για το θέμα αυτό. Uh, uh, Έχω κάποιον άλλον από την ΚΟΕ, όχι. Ράιμον, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ με τη σειρά μου τον εισηγητή, βεβαίως, για την ε, υποβολή του εγγράφου <clears throat> που μπορεί να αποτελέσει καλή βάση. Υπονοεί η έκθεση ότι μόνο η επιβολή του ευρωπαϊκού δικαίου μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση των κρίσεων. Όμως, δεν σημαίνει ότι η εφαρμογή, η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου είναι και η ενδεδειγμένη λύση σε ό,τι αφορά τις πολιτικές. Δεν μπορούμε να δώσουμε δηλαδή και άφεση αμαρτιών για τις χρηματοπιστωτικές πολιτικές των τελευταίων πέντε ετών. Προτιμώ μια πιο ουδέτερη διατύπωση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει και η καλύτερη διαπραγματευτική βάση για μας. Σημαντικές είναι επίσης οι αναφορές σε παραβιάσεις ευρωπαϊκών οδηγιών. Το μεγαλύτερο μέρος των παραβιάσεων αναφέρεται σε φορολογικές, τελωνιακές παραβιάσεις ε, των ε, τελωνιακών δασμών και ούτε καθεξής. Θα τα σημειώσουμε αυτά εμείς σε τροπολογίες μας για, τα τελευταία, για τις τελευταίες τρεις παραγράφους της εκθέσεως. Θα ήθελα να ακούσω στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων περισσότερα επιχειρήματα. Αναφέρομαι στο ενδεχόμενο ίδρυση μια διαρκούς επιτροπής. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής δεν θα ζητάει κάποιος άλλος το λόγο για το Catch Σας ευχαριστώ. Δύο-τρία σχόλια θα ήθελα να κάνω σε σχέση με όσα υπόθηκαν. Καταρχάς ως προς τον σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚ, αγαπητέ φίλε Παύλο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε και να μην αποκαλούμε για το λόγο αυτό τις χώρες με το όνομά τους. Για την έκθεση αυτή διαβάσαμε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απαριθμούνται οι χώρες που δεν συμμορφούνται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οποιοςδήποτε μπορεί να πάει στη διαδικτυακή πύλη, να βρει τη σχετική ιστοσελίδα και να βρει αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι δημόσια, σε πλήρη διαφάνεια. Πριν από τρία χρόνια ήμουν εισηγητής για την έκθεση για τον ανταγωνισμό και είχα τότε τον ίδιο φόβο. Για πρώτη φορά βάλαμε το όνομα της Google ως μια εταιρεία ξεκάθαρα ε, με συμπεριφορά αντιτράστα. Και τελικά 600 ε, ευρωβουλευτές υπερψήφισαν το κείμενο της έκθεσης ανταγωνισμού το οποίο καλούσαμε επιτακτικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσει ενδυνάμει συμπεριφορά αντιτράστα ε, της Google. Για πρώτη φορά λοιπόν δια... διεράγει θα έλεγα αυτή, αυτή η συνένεση, η συγκατάθεση ότι δεν είναι πολιτικός ορθό να ονοματίζουμε συγκεκριμένες εταιρείες ή να ονοματίζουμε συγκεκριμένες χώρες. Όμως οι πολίτες απαιτούν από εμά να μιλούμε ξεκάθαρα για τα ζητήματα, να αρθρώνουμε καθαρό πολιτικό λόγο και όλα αυτά είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οφείλουμε να λύσουμε αυτό το βασικό ζήτημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να προχωρούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με αποκλήσεις στις συμπεριφορές, στις πρακτικές των κρατών μελών. Π.χ. η Δανία, για παράδειγμα, ενδεχομένω έχει την καλύτερη αγορά απασχόληση στον κόσμο και σε κάποιες χώρες στο νότο της Ευρώπης είναι η, χειρότερα, χειρότερη αγορά απασχόλησης στον ανεπτυγμένο κόσμο. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή να ονοματίζουμε τα καλά ξεκάθαρα και τα κακά όχι. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μια ένωση βέλτιστων πρακτικών κατά την άποψή μου οι, χώρες με την καλύτερη νομοθεσία στο εκάστοτε πεδίο να τη βάζουν αυτή την νομοθεσία επιτάπητος και να τη μοιράζονται με άλλες χώρες. Και γι' αυτό ένα σαφές και πολύ σημαντικό ζήτημα είναι να σταματήσει επιτέλους αυτή η συνήθεια ένα νομοθετικό καθεστώς αλλά που ε, παραγγέλνει κανείς και καταναλώνει δωρεάν κατά πώς τον ε, βολεύει. Τελικά αυτά θα τα υπερψηφίσετε ή θα τα καταψηφίσετε. Όμως, θυμάμαι πολύ καλά, Πάμπλο, αυτό που είπατε. Είναι ανάγκη να μην είμαστε συγκεκριμένοι. Σας λέω, το φόβο αυτό τον είχαμε και πριν από τρία χρόνια στην έκθεση ανταγωνισμού, ότι αν πούμε συγκεκριμένο όνομα συγκεκριμένης εταιρεία, δηλαδή της Google, δεν θα τύχει στήριξη η έκθεση. Όμως το βάλαμε, τολμήσαμε να το βάλουμε το όνομα της Google και 600 βουλευτές και πάνω υπερθεμάτισαν και ενέκριναν την έκθεση. Βεβαίως τα πρόθεσμα, οι καθυστερούμενες πληρωμές είναι πράγματα πολύ σημαντικά πριν από τρία χρόνια ε, ξεκίνησε η συζήτηση του θέματος. Πέρσι εγκρίναμε κανονισμό για όλα αυτά. Βάση κάθε οικονομικού συστήματος είναι η Late Payment Directive. Όπως λένε και οι Αμερικάνοι, business κάνουμε μόνο όταν υπάρχει εκταμίευση τελικά. Τότε θεωρούμε ότι έχει κλείσει το business, έχει κλείσει η συμφωνία. Ε, υπάρχει μια επιστολή που λέει ότι αγαπητέ ε, Τζον, μιλάτε για το δυτικό πολιτισμό. Θα έπρεπε να μιλάτε για τη δυνατότητα δυτικού πολιτισμού εάν τηρούνται οι συμφάσεις, αν οι συμφάσεις και αν πληρώνονται οι λογαριασμοί. Είναι γνωστή αυτή η ρίση στο διεθνές στερέωμα Χθες στην Εξπανσιόν, μια ισπανική εφημερίδα, πολύ γνωστή ευρείας κυκλοφορίας, στο σημείωμα του εκδότη ε, ζητούνται, αναφέρονται κυρώσεις ενδεχομένως που η Κομισιόν θα επιβάλλει στο Ισπανικό κράτος λόγω της κακής εφαρμογής της οδηγίας ε, για τις καθυστερούμενες οφειλές και την πληρωμή τους. Στρέφουμε προς τους πράσινους και προς την ΚΟΕ για να πω τα εξής. Ενδεχομένως οι καταληκτικές προθεσμίες δεν ήταν ρεαλιστικές για την ομοθέσια για τα τραπεζικά. Οι πολίτες όμως αυτή την πληροφόρηση δεν την έχουν. Επομένως, θα πρέπει την επόμενη φορά που θα νομοθετήσουμε να είμαστε πολύ πιο ρεαλιστές. Και δεν ζητώ τη δημιουργία της υποεπιτροπής για τη δημιουργία επιπρόσθετης γραφειοκρατίας. Η Σάλη με βοήθησε ιδιαίτερο σε όλη αυτή τη δουλειά. Αναφέρομαι στη δυνατότητα σύστασης μιας υποεπιτροπής ακριβώς για να τονίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Βεβαίως θα το συζητήσουμε, είμαι ανοιχτό ε, σε απόψεις. Δεν είναι και εύκολο να συσταθεί μια επιτροπή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας τρόπος να πούμε στους πολίτες ότι δεν είναι πλέον αποδεκτή η άποψη business as usual, ότι θα είναι συνήθις πρακτική των επιχειρήσεων αυτή. Δεν επιτρέπεται πλέον. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να έχουμε συνένεση και συγκατάθεση ε, και συνεργασία τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Καταλεκτική προεθεσμία για υποβολή τροπολογιών 22 Μαρτίου το μεσημέρι. Εξέταση τροπολογιών 19 Απριλίου. Ψήφιση στην Επιτροπή μας 25-26 Απριλίου. Ψήφιση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 24 Μαΐου. Προχωρούμε στο, στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, κοινό σύστημα φόρου τη θέμενης αξίας όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού η Εισηγητής ο κύριος Σίμων. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε σήμερα στην ψηφοφορία για την έκθεσή μου για την παράταση του ελάχιστου κανονικού συντελεστή του 15% για άλλα δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι τέλος του 2017. Πρόκειται για την τροποποίηση της οδηγίας περί, προ, περί φόρου αξίας, που επειδή είναι οδηγία του Συμβουλίου, προβλέπει γνωμοδότηση μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κανόνας ότι ο ελάχιστος συντελεστής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15% ήδη έχει ε, το. 1993 και έχει μέχρι τώρα παραταθεί κατά πέντε, ε, φορές. Μιλούμε για μια ενιαία αγορά η οποία δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Δεν προχωρούμε σε εναρμόνιση των φορολογιών. Παρόλα αυτά αναμέναμε μία λύση η οποία δεν έχει δοθεί ως τώρα. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να αναφέρω θετικά ότι με το VAT Action Plan της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα δημοσιευθεί την επόμενη Τετάρτη 23 Μαρτίου, γίνεται άλλη μια προσπάθεια από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εισαχθεί ένα τελεσίδικο πλέον, ένα οριστικό σύστημα φόρου προσθεμένης αξίας, με στόχο την καταπολέμηση των φοροαπατών γύρω από τον ΦΠΑ. Και σύμφωνα και με την έκθεση ε, του ε, συναδέλφου μας Βέρνερ Λάγκεν για το θέμα του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή, συντελεστή ΦΠΑ δηλαδή, αρχίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάλι μια νέα συζήτηση. Στους επόμενους μήνες θα πρέπει να ξεκαθαριστεί εάν οι χώρες μέλη επιθυμούν την διατήρηση του φορολογικού αυτού συντελεστή ή εάν προτιμούν ένα εύκαμπτο σύστημα το οποίο δεν θα περιλαμβάνει φορολογικό συντελεστή. Επειδή η συζήτηση αυτή οφείλει να γίνει και μάλιστα επίκαιρα, είναι συνεπές ότι η παράταση του ελάχιστου συντελεστή ΦΠΑ που συζητούμε σήμερα, η παράταση λοιπόν θα πρέπει να ισχύσει μονάχα για μια διετία. Ωστόσο, μια κριτική παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με καθυστέρηση τη σχετική πρόταση, ώστε να καθίσταται απαραίτητη μια αναδρομική εφαρμογή από 1η 2016 Όπως εξήγησε η κυρία Πάρνουβα αλλά και ο Βέρνε Λάγκεν, δεν είναι ξεκάθαρη αυτή η διαδικασία, όσο και να προσπαθήσει και να την ευρωποιήσει. Δεν είναι καλή Θεωρώ πάντως ότι σήμερα πρέπει να υπερψηφίσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα όμως, εν προκειμένου, να πω και πάλι, ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένουμε περισσότερο πρόσωσχεδιασμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, Ευχαριστώ από το ΕΛΚ, Εύα Παουνόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, όπως ήδη έχετε ενημερωθεί. Η ομάδα μας είναι κατά της ε, ε, απλουστευμένης διαδικασίας. Θέλουμε να είναι ανοιχτή αυτή η πρόταση στις για Και εμείς είμαστε κατά αυτού γιατί η Επιτροπή καθυστέρησε στην υποβολή των τροπολογιών στην οδηγία. Οι τρέχοντες κανόνες ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015 και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει νομοθεσία για δύο ολόκληρους μήνες για το ελάχιστο κατόφλι του ΦΠΑ και γι' αυτό προτείναμε αυτή την τροπολογία διότι πιστεύουμε δηλαδή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να θεωρήσει την Επιτροπή υπόλογη και θα ήθελα να σας ζητήσω να στηρίξετε την τροπολογία υπαριθμών 1, η οποία όπως είπε και ο εισηγητής υπογραμμίζει το γεγονός ότι θεωρούμε θλιβερό το γεγονός ότι η Επιτροπή καθυστέρησε να υποβάλει την πρόταση και έτσι είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή του κατώτατου συντελεστή και η θέση σε ισχύ της διάρκειας της υποχρέωσης αυτής. Πρέπει να υπάρχει συνοχή στην ε, νομοθεσία, να μην υπάρχει νομοθετικό κενό χρονικά και στην τροπολογία 5 για την οποία θέλουμε τη στήριξή σας θέλουμε η διάρκεια της υποχρέωσης να εκτείνεται στα 5 χρόνια και όχι στα 2 η η Επιτροπή θεωρεί ότι θα υπάρχει ένα νέο σύστημα ΦΠΑ μέχρι το 2018, όμως εμείς πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι κανόνες να είναι ε, ίδιοι και να ισχύσουν για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, ε, ειδικότερα εάν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει καθυστέρηση στην μελλοντική νομοθετική διαδικασία. Συμφωνώ, πρέπει να εξυγχρονιστεί το τρέχον σύστημα ΦΠΑ για να μην υπάρχουν κενά που ξεπερνούν τα 170 δις ευρώ αυτή τη στιγμή, οι αποκλήσεις στο ΦΠΑ δηλαδή. Και άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις προκλήσεις, τις καινοτομίες στο ψηφιακό περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει, οι κανόνες που ισχύουν για τους συντελεστές ΦΠΑ θα πρέπει να εφαρμόζονται για να μειωθεί και η απόκληση ε, των συντελεστών. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές υπάρχει κάποιος που θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Υπενθυμίζω τα όσα είπα στην τελευταία φορά που το συζητήσαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ε, σχετικό σχεδιασμό. Ε, εύχομαι να πάει καλά. Θα περιοριστώ μόνο στο σχόλιο σήμερα ότι έχουμε αναγνώσει τις τροπολογίες του Λαϊκού Κόμματος. Ε, Ευχαρίστω να τις υποστηρίξουμε. Κάποιες προτάσεις είναι καλές και όπως είπα μας βρίσκουν σύμφωνος. ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Σας ευχαριστώ. Πέτρ Γέτσεκ. Σας ευχαριστώ. Η αλλαγή αυτή που προτείνεται θα πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά μέσα στα πλαίσια και του σχεδίου δράσεως που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. εγώ νομίζω ότι είναι πρόημη μια οποιαδήποτε παρατεταμένη παράταση, ας το πω έτσι, του ελάχιστου συντελεστή ΦΠΑ. Είναι λυπηρό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την παράταση του ελάχιστου συντελεστή με καθυστέρηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Ματίας, όχι. Ενωτική αριστερά, όχι. Κανείς ε, για την Ευρωπαϊκή Ερνοτική Αριστερά. Ο κ. Σουρτασούν ούτε. Καλώς η Κομισιόν νεύει αποφατικά. Κύριε Σιγητά, αγαπητές και αγαπητοί, ευχαριστώ για τις σημαντικές αυτές παρεμβάσεις. Κυρία Πάουνοβα, μπορεί βεβαίως να υποστηρίξει και τις δύο πλευρές ε, το χρονικό σχεδιασμό και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ας είμαστε όμως πιο φιλόδοξοι. Ως εισηγητής θεωρώ ότι εάν έχουμε ένα χρονικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε ενδεχομένω σε μια οριστική λύση, να μην ταχθούμε υπέρ κάποιων λύσεων που ενδεχομένω να αντιβαίνουν την ε, στην προσπάθεια αυτή. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω ε, πλήρω το νόημα των επιχειρημάτων σα. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Μπορούμε να προχωρήσουμε εμείς στην ψηφοφορία. Γιατί λίγο έχουμε καθυστερήσει. Σε δύο λεπτά λοιπόν, ψηφοφορία κυρίε και κύριοι. Παρακαλώ να βάλετε τις ε, κάρτες ψηφοφορία στην σχισμή του μηχανήματος. are perfectly in time. We're supposed to be 11, 10 past 11. Είμαστε απολύτως εντάξει σχετικά με το χρόνο, λέει ο Πρόεδρος. Είναι 12, 11, 11 η ώρα και 12 λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ, ας κάνουμε πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Test, test, still open for the... Πρόκειται για δοκιμαστική ψηφοφορία ακόμη. Gunnar, put the card. We wait for... Βάλτε την κάρτα σας, Gunnar. Περιμένουμε. Ωραία. Πέρα τη ψηφοφορία, θαυμάσια λοιπόν, μπορούμε να αρχίσουμε την πραγματική ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει για την 5 Πέρας. Απερίφθη. Υπαριθμών 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Α, με συγχωρείτε, δεν είπα τις αποχές. Όχι, check, λέει ο πρόεδρος, επαλήθευση. Πέρας. Μάλιστα εγκρίνεται. υπαριθμόν 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. υπαριθμόν 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή ψήφος επί του τροποποιηθέντος κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. 37 υπέρ, 5 κατά και 4 αποχές. Ψήφισμα, ε, μάλλον ε, νομοθετικού περιεχομένου ψήφισμα. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Ας περιμένουμε λίγο για να ψηφίσουν όλοι. Σύντομα παρακαλώ. Ωραία, ψηφίσατε και εσείς. Πέρας. 41 ψήφοι υπέρ, 5 κατά και 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται στις 22 Μαρτίου στις 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ και εδώ λίγη συνεδρίαση.